I think we can start. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, κυρίως διότι ο κυρίος Παντεκάμ με ρώτησε πότε θα ξεκινήσουμε. Με 10 λεπτά καθυστέρηση, επομένως είναι καλή ώρα να ξεκινήσουμε. Καταρχάς αποφάσεις των, συντονισμών, ε, των συντονιστών, συγγνώμη, τις ε, έχουμε διανύμει. Αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι τις 6.30 κατά τη λήξη της συνεδρίασης, ε, θεωρείτε ότι έχουν εγκριθεί. Διαβάστε λοιπόν προσεκτικά και πείτε μας αν υπάρχει κάποιο λάθος. Πολύ ωραία. Δεύτερη ανακοίνωση. Είχαμε τους συντονιστές. Ο Πίτερ Μπάλλας δεν θα είναι παρόν διότι ακυρώθηκε η πτήση του. Θα δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε την ημερήσια διάταξη για να μην χρειαστεί να περιμένουμε. Κατόπιν ε, έχουμε παρουσίαση μελέτης σχετικά με την κοινωνική ένταξη στον τομέα των ε, δημόσιων μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζω λοιπόν ε, τους κυρίους που θα μας κάνουν την παρουσίαση. Κυρία Λουντοβίτσι, έχετε πρώτη τον λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Okay. Okay. Uh, many thanks for... Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να σας κάνω αυτή την παρουσίαση των μελετών που κάναμε εξ ονόματος της Επιτροπής Δημόσιας Μεταφοράς και Κοινωνικής Συμπερίληψης, ένταξης. Είναι νέο το ζήτημα αυτό, γιατί όταν μιλούμε για τις δημόσιες μεταφορές, συνήθως λίγη προσοχή δίδεται σε θέματα κοινωνικής ένταξης ή συμπερίληψης. Αυτό το οποίο κάναμε εδώ είναι το εξής. Προσπαθούμε να κάνουμε μια επισκόπηση του πώς συνδέεται η κοινωνική ένταξη με τις δημόσιες μεταφορές, ε, αναθεωρώντας, εξετάζοντας τη βιβλιογραφία και ορισμένα εμπειρικά στοιχεία. Τώρα, ε, αναγνωρίζεται όλο και πιο ευρέως το γεγονός ότι για να ε, καταπολεμηθεί η φτώχεια και να μειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, για, ειδικά για ορισμένες μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες, οι δημόσιες μεταφορές έχουν ένα ρόλο καθοριστικό ε, να ε, διαδραματίσουν. Μπορούμε να έχουμε παραδείγματα πολιτικών και ε, πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Και τα έχουμε αυτά. Και στο τέλος της παρουσίασής μας της μελέτης μας υπογραμμίζουμε ορισμένα ζητήματα που αξίζει να μελετηθούν περαιτέρω. Υπογραμμίζουμε τον ενδυνάμει ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράδειγμα, διότι μπορούν να αυξήσουν την προσοχή που δίδεται στο ρόλο των δημοσίων μεταφορών ως καταλήτης για περισσότερη κοινωνική ένταξη. Συζητούμε στη μελέτη μας τι σημαίνει ο όρος κοινωνική ένταξη Υπάρχει πολύ εκτενής βιβλιογραφία για το θέμα αυτό, δεν θα ε, εμβαθύνω, ωστόσο, σήμερα και τώρα, ωστόσο θέλω να τονίσω ότι η κοινωνική ένταξη είναι ένα μια πολυδιάστατη έννοια. Σημαίνει τη δυνατότητα που έχει κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως του φίλου του, της φιλής του, της ηλικία του, του εισοδήματός του, της κατάστασής του να συμμετέχει στην κοινωνική και πολιτική ε, και οικονομική ζωή. Είναι η δυνατότητα πρόσβαση στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Να σας δώσω κάποια στοιχεία για το πώς οι άνθρωποι στην Ευρώπη βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Λαμβάνοντας υπόψη έναν από τους δείκτες κοινωνικού αποκλεισμού που είναι ο κίνδυνος φτώχειας. Το 2013 περίπου ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη είναι φτωχοί. Θεωρούνται φτωχοί. Ένα στους τέσσερις στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτό. Άρα ε, ότι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και ε, κοινωνικού αποκλεισμού. Μιλάμε για 123 εκατομμύρια ανθρώπους. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και με την κρίση αυτό το, αυτός ο αριθμός αυξάνεται. Οι πιο μειονεκτικές, ε, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ε, αντιμετωπίζουν περισσότερο αυτό το κίνδυνο. Και βλέπουμε τα στοιχεία από το 2009 μέχρι το 2013 σημειώθηκε αύξηση, προστέθηκαν 7 εκατομμύρια άνθρωποι στο συνολικό αριθμό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο της φτώχειας. Βεβαίως οι διαφορές είναι πλήστες μεταξύ των χωρών. Και αυτό δείχνει τη διαφορά των ε, συστημάτων κράτους πρόνοιας που έχει κάθε χώρα, ε, ε, τη διαφορά στην προσπάθεια πολιτικής που εφαρμόζει κάθε χώρα για να προσεγγίσει το θέμα αυτό. Αλλά οφείλονται βέβαια διαφορές και στις μεγάλες διαφορές των οικονομικών συνθήκων. Οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, είναι οι χώρες που βίωσαν και τη μεγαλύτερη αύξηση του κινδύνου φτώχειας. Δεν ξέρω αν βλέπετε αρκετά καλά σε αυτή την οθόνη που είναι απομακρυσμένη. Εδώ έχουμε μια γραφική παράσταση, ένα γράφημα ε, που παρουσιάζονται οι πληθυσμοί ανά χώρα που κινδυνεύουν με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Στην κόκκινη λωρίδα είναι ο ευρωπαϊκός μέσος 24,8% του πληθυσμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά Μεσοόρο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά πιο υψηλό στη Βουλγαρία 49%, Ρουμανία 42%, Ελλάδα σχεδόν 35% και ούτω καθεξής, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει κατά πολύ συγκριτικά με το μέσο όρο σε χώρες όπως οι κάτω χώρες 15%, η Σουηδία 15,6%, η η Τσεχία και ούτω καθεξής. Άρα πολύ μεγάλες διαφορές παραμένουν μεταξύ των χωρών. Ποιοι είναι τώρα οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Εάν κάποιος δηλαδή έχει απασχόληση, έχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα ή όχι. Υπάρχουν παράγοντες που σχετίζονται με το επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την απασχολησιμότητα των ατόμων. Όσο πιο μορφωμένα είναι τα άτομα, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν να έχουν απασχόληση και μάλιστα με ικανοποιητικές απολαβές. Άλλος παράγοντας είναι η σύνθεση του νοικοκυριού, ε, του σπιτιού δηλαδή, της οικογένειας και το κατά πόσο ζει σε αστικές περιοχές ή στην Ήπεθρο. Εκτός από αυτούς τους γενικούς παράγοντες που προανέφερα, υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυξάνουν το κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Όπως για παράδειγμα το να είναι κανείς άτομο με αναπηρία, να έχει υπόβαθρο μετανάστη, να ανήκει σε μια μειονοτική εθνοτική ομάδα, να είναι γυναίκα γιατί οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχεια σε σχέση με τους άνδρες. Να έχει χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και χαμηλή εκπαίδευση, παύλα μόρφωση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λειτουργούν αθρηστικά. Υπάρχουν ας πούμε γυναίκες με ε, καταγωγή μετανάστη, με χαμηλό ε, επίπεδο εκπαίδευσης που διαβιούν στην Ήπεθρο. Είναι πολυδιάστατη η μορφή του κοινωνικού τους αποκλεισμού και φυσικά έχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό το γράφημα, άλλωστε να πω παρεθετικά ότι όλα τα αριθμητικά στοιχεία, τα νούμερα τα βλέπετε στην έκθεση, μπορείτε να τα βρείτε ε, η οποία έχει αναρτηθεί και στο διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν το γράφημα, αυτή η γραφική παράσταση μας δείχνει τον κίνδυνο φτώχειας για διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού. Είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος φτώχειας των ανέργων. Το 67% των ανέργων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, γιατί δεν έχουν εισόδημα. Τα παιδιά και κυρίως τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ή τα παιδιά ανέργων έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο φτώχειας. Οι μετανάστες, όσοι έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και όσοι ζουν σε, σε περιοχές που δεν υπάρχει μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα. Βλέπετε, αυτοί αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχεια. Βλέπετε ότι δεν έχουμε αναφορά σε ε, ε αν όμως μπούμε σε τέτοιου είδους πληθυσμιακές ομάδες, αν δηλαδή εμβαθύνουμε ε, στις ε, πληθυσμιακές ομάδες της τρίτης ηλικίας και των ατόμων με αναπηρία, ε, να δούμε ποιες περαιτέρω δυσκολίες αντιμετωπίζουν αυτές οι κοινωνικές ομάδες, βλέπουμε ότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος ε, να έχει κανείς μια ανεξάρτητη ζωή. Αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες είναι πολύ πιο ευπαθείς στον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι ηλικιωμένοι δηλαδή και τα άτομα με αναπηρίες. Επομένως, οι δημόσιες μεταφορές μπορούν να στηρίξουν την κοινωνική ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Και αν ε, αυτά τα θέματα δεν τα λάβει υπόψη της η πολιτική για τις μεταφορές, τότε η πολιτική μεταφορών από μόνη της αυξάνει τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Πρέπει κανείς να έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, σε ευκαιρίες απασχόλησης, σε καλύτερες κοινωνικές σχέσεις και σε μείωση της κοινωνικής απομόνωσης. Οι ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες, τα παιδιά ανέργων ή ατόμων χαμηλού μορφωτικού επίπεδου μεταναστών κτλ. Αυτοί βρίσκονται σε ακόμα πιο μειονεκτική θέση γιατί αυτοί ακριβώς είναι που χρησιμοποιούν τις δημόσιες μεταφορές πολύ περισσότερο από ό,τι οποιοδήποτε άλλος, γιατί αυτοί είναι που κατεξοχήν δεν έχουν όχημα ιδιωτικό, ε, γιοταχή ή δεν έχουν χρήματα αρκετά για να επιλέξουν άλλους τρόπους μεταφοράς. Επίσης, ο αρνητικός αντίκτυπος του, αντίκτυπος του συστήματος μεταφορών στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία κτλ. Ε, θα ε, επηρεάσει αυτές ακριβώς τις κοινωνικές ομάδες πολύ περισσότερο από ό,τι τις άλλες. Δεν θα, τώρα θα σας αναλύσω όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία που βλέπετε στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Ε, είναι όμως ενδιαφέροντα γιατί τα έχουμε βρει από την επιστημονική βιβλιογραφία. Είναι απολύτως έγκυρα και δείχνουν το φαύλο κύκλο που δημιουργείται με αυτή την αλληλεπίδραση με μεταξύ του κοινωνικού αποκλεισμού, του αποκλεισμού από τις δημόσιες μεταφορές και των συστημάτων κινητικότητας. Αυτά τα τρία αλληλεπιδρούν. Όσοι είναι κοινωνικώς αποκλεισμένοι δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια μέσα μεταφοράς και αν τα δημόσια μέσα μεταφοράς δεν στηρίξουν αυτά τα άτομα για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, σε θέσεις απασχόλησης, σε κοινωνική δικτύωση, τότε τα μειονεκτικά στοιχεία αυτών των ατόμων και τα προβλήματά τους, η μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται, γίνεται, ε, επιδεινώνεται, γίνεται ακόμα πιο σοβαρή. Το είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι διαφέρει αναλόγως με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν και διαφέρει επίσης και αναλόγως με το για ποια ομάδα μιλάμε. Για παράδειγμα, για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ανεπηρίες ε, το βασικό πρόβλημα είναι η προσβασιμότητα η σωματική. Ε, δηλαδή πώς μπορεί κανείς να ανέβει στο δημόσιο λεωφορείο, να πάρει, να μετακινηθεί από την αποβάθρα και να μπει μέσα στο βαγόνι του ε, σιδηρόδρομου, του τρένου. Επίσης, πρόβλημα είναι η πληροφόρηση για τα χρονοδιαγράμματα, για τα ωράρια, για τις τιμές και το καθεξής. Ενώ, για παράδειγμα, για τις γυναίκες το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι η ασφάλεια. Δηλαδή να μπορούν οι γυναίκες ακόμα και το βράδυ να παίρνουν τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα για τις γυναίκες είναι το γεγονός ότι Σύμφωνα με πάρα πολλές μελέτες, ενώ οι άνδρες χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς κυρίως κατά τις ώρες εχμής για να πάνε στη δουλειά, δηλαδή απ' έξω προς το κέντρο των πόλεων ή αντιστρόφως, για τις γυναίκες δε το είδος κινητικότητας διαφέρει. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς σε διάφορα ωράρια, σε διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί δεν χρησιμοποιούν μόνο τα μέσα μεταφοράς στα δημόσια για να πάνε στη δουλειά τους, αλλά και για να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο ή να συνοδεύσουν τα ηλικιωμένα μέλη της ευρύτερης οικογένειας στις υπηρεσίες υγείας ή για να ε, πάνε για ψώνια και Άρα η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς από τις γυναίκες είναι τελείως διαφορετική από αυτή που κάνουν οι άνδρες. Και είναι σημαντικό να λάβει κανείς υπόψη του αυτό το ζήτημα όταν σχεδιάζει στρατηγικές μεταφορών. Γιατί ο συνήθις τρόπος δημόσιας μεταφοράς, του να έχει δηλαδή κανείς ένα σωρό συχνά, πώς να το πω, ε, δρομολόγια λεωφορείου και μετρό και τρένων κατά τις ώρες ε, εχμής αυτό είναι το παραδοσιακό. Αυτό, όμως αυτό συμφέρει και είναι καλό για τους άνδρες, αλλά όχι τόσο για τις γυναίκες. Οι γυναίκες χρειάζονται ένα περισσότερο ε, κατανεμημένο χρονοδιάγραμμα δρομολογίων π.χ. καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και κυρίως να, ε, καλύτερη σχεδίαση της ενδομεταφοράς στην, ε, στο προάστιο, στο διαμέρισμα, το δημοτικό ε, του καθενός. Συνήθως θέλει κανείς να πάει στις κοινωνικές υπηρεσίες ε, που είναι ε, πιο κοντά του γεωγραφικά και θέλει να το κάνει αυτό εκτός ορών, ορών εχμής. Ποιες είναι οι πρόσφατες εξελίξεις. ως προς την ανάπτυξη της πολιτικής. Λοιπόν, το τελευταίο χρόνο ε, γίνεται όλο και πιο συνειδητή αυτή η ανάγκη ε, του ότι οι δημόσιες μεταφορές πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. Το, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής εμπλέκονται εκεί. Μιλούμε για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών μεταξύ άλλων. Αυτά τα ζητήματα έχουν απασχολήσει τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ένα ε, σημαντικό θέμα είναι ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν τοπικά έργα, τοπικές πολιτικές, ε, για να στηρίξουν πιλωτικά προγράμματα που στόχευαν στην κάλυψη των αναγκών αυτών των πληθυσμιακών ομάδων των ευπαθών. Οι πιο ενδιαφέρουσες καλές ε, πρακτικές, τα πιο ενδιαφέροντα έργα που έχουν εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο, χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής. Τώρα, τα εμπειρικά στοιχεία δεν έχω χρόνο να σας τα παρουσιάσω ενδελεχώς κάνουμε ανάλυση ανά ομάδες στόχους και δείχνουμε ποιες είναι οι βασικές ανάγκες, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι ε, κοινωνικές ομάδες στην πρόσβαση ε, στις δημόσιες μεταφορές και ε, αναλύουμε εμπειρικά τα στοιχεία που υπάρχουν για το πώς εφαρμόστηκε σε τοπικό επίπεδο η εκάστοτε πολιτική για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Για παράδειγμα, δημόσιες μεταφορές από το σπίτι στο σχολείο για νέους ανθρώπους, για φοιτητές και μαθητές, για να βελτιωθεί η ασφάλεια του τρόπου μεταφοράς των παιδιών, για να προωθηθεί η χρήση των δημόσιων μέσων ε, μεταφοράς το βράδυ από τους νέους, κυρίως την Παρασκευή το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ και να χρησιμοποιηθεί νέα τεχνολογία για να αναπτυχθούν νέα είδη μεταφοράς. Αυτό μας έχει ενδιαφέρα. Ε, μας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν ξέρετε το Black Current ε, χρησιμοποιείται πολύ από τους νέους, βασίζεται στη τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, παρέχονται υπηρεσίες από ιδιωτικούς φορείς και ήθελα να το αναφέρω γιατί είναι σημαντικό. Τώρα, για τους ηλικιωμένους, για την τρίτη ηλικία. Μεταφορά ευέλικτη, πόρτα-πόρτα, με ταξί, με εθελοντές μη κυβερνητικών οργανώσεων που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης σημειώνεται αύξηση στην παροχή υπηρεσιών πόρτα-πόρτα και κατόπιν αιτήματος on demand, αναλόγως δηλαδή με τη ζήτηση του που έχει ο ηλικιωμένος ή το άτομο με αναπηρίες. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις δύο πληθυσμιακές ομάδες αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν. Όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται η τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας για να αρθούν οι φραγμοί Τελειώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι και για τις γυναίκες το ίδιο ισχύει. Ε, δόθηκε έμφαση σε μέτρα ασφαλείας για να, δι... να βελτιωθεί η δυνατότητα των γυναικών να μπορούν να ταξιδεύουν το βράδυ με ασφάλεια. Και άλλαξε ο σχεδιασμός η παρουσίαση των τρόπων μεταφοράς για να στηρίξει τις γυναίκες που έχουν παιδιά μαζί τους ή που συνοδεύουν ηλικιωμένους. Για παράδειγμα, πριν από λίγους μήνες πήγα στη Μαδρίτη και είδα ότι στα λεωφορεία υπάρχει συγκεκριμένη θέση για μητέρες με πολύ μικρά παιδιά. Όπου <clears throat> μπορεί κανείς να βάλει το παιδί σε ένα καθίσμα ασφαλείας τελικά. Δεν θα σας πω τι ακριβώς γίνεται για τους ανέργους και για τα άτομα χαμηλού εισοδήματος γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Το ίδιο είναι όμως το ζήτημα. Συγκεκριμένες υπηρεσίες να παρέχονται που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των μειονεκτικών ομάδων. Για παράδειγμα, για τους μετανάστες ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η γλώσσα. Επομένως, η παροχή πληροφοριών με διαφορετικές γλώσσες για να ξέρει κανείς και να καταλαβαίνει ε, τι είδους μέσο μεταφοράς διατίθεται είναι κάτι το σημαντικό. Ένα άλλο θέμα είναι όσοι ζουν στην Ήπεθρο και είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό γιατί με τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες λόγω των πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης, ένα από τα πρώτα μέτρα ήταν να μειωθεί η δημόσια συγκοινωνία σε γεωγραφικές περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Και αυτό πλήττει κυρίως στην τρίτη ηλικία η οποία αποκλείεται όλο και περισσότερο. Άλλωστε η Ήπεθρος κατοικείται κυρίως από ηλικιωμένους. Οι νέοι εγκαταλείπουν την Ήπεθρο. Μεγάλο ζήτημα αυτό λοιπόν. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματικότητα με την απόφ και την πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την αποτελεσματικότητα και την, ε, τις περικοπές στις δημόσιες με την ισονομία για όλους. Στο μέλλον λοιπόν οι προκλήσεις των δημόσιων μέσων μεταφοράς ε, από πλευράς κοινωνικού αποκλεισμού θα αυξηθούν. Γιατί το πρόβλημα γύρανσης, πληθυσμιακής γύρανσης της Ευρώπης θα οξύνεται. Άρα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα κινητικότητας των ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες. Και πολύ μεγαλύτερη είναι η συχνότητα των μεταναστευτικών ροών και η κινητικότητα εντός Ευρώπης των ατόμων που αλλάζουν χώρα για να βρουν θέσεις απασχόλησης μεταξύ άλλων. Και αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ληφθούν υπόψη αυτά τα θέματα. Υπάρχει πρόβλημα με τις αυξημένες ανισορροπίες από πλευράς πληθυσμιακής. Δηλαδή, οι αστικές περιοχές πλήττονται από συμφόρηση κυκλοφοριακή και έντονη πληθυσμιακή πυκνότητα, ενώ η ύπεθρος πλήττεται από την εγκατάλειψη, από την ερήμωση αυτής και πρέπει να λυθούν αυτά τα θέματα. Στο μέλλον θα είναι σημαντικό να λύσει κανείς τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, να θεωρήσει ότι υπάρχει ζήτημα κοινωνικού αποκλεισμού ε, σε κάθε πολιτική για τις δημόσιες μεταφορές που ε, εφαρμόζει, γιατί είναι σημαντικό ε, κομμάτι, σημαντικό σκέλος. Δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Αν το θέμα είναι να, κόψουμε, να περικόψουμε το κόστος, ε, τότε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις νέες τεχνολογίες και να μάθουμε περισσότερα για αυτά τα πιλωτικά προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονται από κάτω προς τα πάνω. Για το κατά πόσο μπορούμε να παραδειγματιστούμε για το τι πρέπει να κάνουμε. Και τρίτον, πρέπει να εμπλέξουμε όλο και περισσότερο τους ιδιωτικούς ε, παρόχους μεταφοράς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τον τριτογενή τομέα της ε, οικονομίας, των μη κυβερ... τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την κοινωνική πολιτική. Μπορούν εκείνοι να δίνουν κάποιες δυνατότητες μεταφοράς σε ε, κοινωνικές ομάδες ευπαθείς. Έχουμε το παράδειγμα των ονοχημάτων, των αυτοκινήτων μπλα μπλα. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Μοιραζόμαστε τις ανάγκες μας, ταιριάζουμε τις ανάγκες του ενός με τις ανάγκες του, του άλλου. Δεν χρειάζεται δηλαδή δημόσια παρέμβαση και άρα δεν χρειάζονται δημόσια δαπάνες. Ωστόσο σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση. Συμφωνώ απολύτως. Γίνεται εδώ ανάλυση των ομάδων υψηλού κινδύνου, των ομάδων δηλαδή εις βάρος των οποίων ε, γίνονται, μάλλον που αποκλείονται από την κοινωνία. Αυτοί οι αποκλεισμένοι είναι ακριβώς τα άτομα με αναπηρίες, ε, οι μετανάστες, οι άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα, οι άνεργοι. και τα άτομα που ζουν σε υπαίθριες περιοχές που απέχουν πολύ από αστικές περιοχές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στις πόλεις δεν υπάρχουν αποκλεισμένοι κοινωνικά άνθρωποι και τους οποίους θα πρέπει να εντάξουμε καλύτερα. Η γύρανση του πληθυσμού, ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών, είναι παράγοντες που συμβάλλουν περισσότερο στην εξέλιξη αυτή και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Σημαντικές εδώ είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όταν κάποιος είναι άνεργος, όταν δεν έχει λάβει επαρκή μόρφωση, περιθωριοποιείται. Και αναφέρατε επίσης την ευαισθητοποίηση των δημάρχων, των αρχών, των ανθρώπων που είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη αυτών των μικρών κοινοτήτων. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν δεν υπάρχουν δυνατότητες για τους στοχούς, τους ηλικιωμένους κλπ. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι ήδη φτωχοί, αλλά η κατάστασή τους επιδεινώνεται. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται το κοινωνικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εργαστούμε εδώ σε δύο επίπεδα, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, τις κυβερνήσεις, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει με χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων. θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες κατά την κατανομή των πόρων. Ε, ένας παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη θα πρέπει να είναι ε, αν λαμβάνονται υπόψη οι ε, κοινωνικά αποκλεισμένοι και αν βοηθώνται να ενταχθούν. θα μπορούσαμε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δώσουμε κάποιες συμβουλές, κάποιες οδηγίες, αλλά είναι θέμα που είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο δήμων. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τους ανθρώπους αυτούς. Και κάτι ακόμα όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες και τα εμπόδια που συναντούν. Σημαντικό δεν είναι μόνο το χρηματοδοτικό. Σε πολλά μέρη δεν υπάρχουν υποδομές για άτομα με αναπηρία, δεν μπορούν καν να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία μπορεί να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση αυτή. Είναι θλιβερό ότι σχεδόν το 1 τέταρτο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν ε, τέτοιους κινδύνους και θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Και κάποιος που ε, ε, έχει δουλειά, κινείται με τελείως διαφορετικό τρόπο, έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αυτό τον βοηθάει να πετύχει στη ζωή του. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα. Ξέρω ότι είναι εύκολο να μιλάει κανείς ε, όταν προέρχεται από χώρα που δεν έχει πολλούς μετανάστες όπως είναι η Πολωνία. Αλλά έχω συνομιλήσει με πολλούς μετανάστες οι οποίοι μου έχουν πει ότι αποκλείονται με διτό τρόπο, ζουν σε φτωχές περιοχές, δεν εντάσσονται στην κοινωνία και συχνά όταν προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες δεν έχουν καμία ελπίδα ότι θα αλλάξουν οι συνθήκες διαβίωσής τους. Και τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα κλίμα στο οποίο υπάρχει εντύπωση ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξεφύγουν από την φτώχεια. Θα πρέπει να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κρυσίνη Βοτολό. Σα ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για να μπορέσουν όλοι να μιλήσουν. Καταρχήν να ευχαριστήσω του συντάκτες αυτής της μελέτης που μα επιτρέπει καλύτερα να καταλάβουμε την πραγματικότητα του αντικτύπου των δημόσιων μεταφορών στην καθημερινή ζωή των συμπολιτών μα και να λάβει υπόψη καλύτερα την κοινωνική διάσταση των μεταμεταφορών από την αρχή της θητείας και μάλιστα μέσα στο πλαίσιο των εργασιών για την αναθεώρηση του Λευκού Βιβλίου και της μεταρρύθμισης της αστικής μετακίνησης, θεώρησα ότι ο δημόσιο τομέας θα πρέπει να θεωρηθεί ως <clears throat> ένας βασικός τομέας για να καταπολεμηθεί η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικό αποκλεισμό. Και χαίρομαι που διαβάζω εδώ ότι οι δημόσιε μεταφορέ αποτελούν το μοναδικό τρόπο για να λυθεί το πρόβλημα κινητικότητα ορισμένων ομάδων που είναι κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτε με πάνω από 200 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη που κινδυνεύουν να πέσουν στον κύκλο της κοινωνικού αποκλεισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, τον, να, να ενδυναμώσει τις πολιτικές της. Μόνο το 32% σήμερα των Ευρωπαίων πολιτών χρησιμοποιεί τις δημόσιες μεταφορές μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τα πάει καλύτερα και ελπίζω πως η Κομισιόν θα ιδιοποιηθεί τον στόχο να διπλασιαστεί η χρήση των δημοσίων μεταφορών μέχρι το 2030 μέσα στην αναθεώρηση του Λευκού Βιβλίου. Κάτι που θα πρέπει ίσω περισσότερο να αναπτυχθεί στι συστάσει τη μελέτη είναι η ανάγκη να προωθηθεί η έννοια τη υποχρέωση τη δημόσια υπηρεσία, ώστε ακριβώ να εξασφαλιστεί στους πολίτες μια μη διακριτική ε, πρόσβαση υπό τι καλύτερε δυνατές συνθήκες. Είναι ένα διακύβευμα που δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί και που θα πρέπει να πάρει σημαίνουσα θέση στην αναθεώρηση τη Λευκή Βίβλου. Άνοιγμα δε των ε, συνδρομικών αγορών δεν θα πρέπει να, ορι... να να καταλήξει στις στο να φεθούν οι λιγότερο αποδοτικές γραμμές στους ιδιώτες ε, ε, φορείς. Ε, αυτή η καθολική αποστολή παίζει ρόλο πολύ μεγάλο. Η απελευθέρωση του σιδηροδρόμου δεν θα πρέπει να ε, επιτρέψει τη συγκέντρωση των ροών μεταφορών στα μεγάλα οικονομικά κέντρα και να αφήσει στην μοίρα τους τις πιο, λιγότερο ελκυστικές γραμμές και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Καρίμα Ντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως εισηγήτρια για την αστική κινητικότητα στην Ευρώπη ε, θα πρέπει να σας πω ότι και εσείς τονίζετε αυτά τα κακό κείμενα. Όταν ακούμε δηλαδή τα νούμερα 1 τέταρτο, 1 των Ευρωπαίων πολιτών κινδυνεύει να πέσει μέσα σε μια λέξη στην ε, επισφάλεια της ε, κινητικότητας. 1 τέταρτο του πληθυσμού. Δεν θα μπορεί δηλαδή να μετακινηθεί. Δηλαδή δεν θα μπορεί ούτε να έχει πρόσβαση στην παιδεία, ούτε στην ψυχαγωγία, ούτε στην εργασία και σε έναν άλλο μακρύ κατάλογο πραγμάτων. Πιστεύω πως είναι μια πληγή αυτή που δεν έχουμε το δικαίωμα να την ε, αγνοήσουμε. Είπατε πριν από λίγο πως η τεχνολογία θα βοηθήσει, θα προσπαθήσει κάπως να βοηθήσει ώστε τα πιο ευάλωτα άτομα να έχουν πρόσβαση στην κινητικότητα. Όμως πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Γιατί ακόμα και για τα αυτοκίνητα εκείνα, τα... Ε, οι περισσότεροι και οι πιο φτωχοί δεν έχουν πρόσβαση στα εφή τηλέφωνα, στα smartphone. Αυτά τα μέσα λοιπόν ε, ε, δεν είναι πάντοτε προσιτά στους φτωχότερους. Πολλοί δεν έχουν καν πρόσβαση στο ίντερνετ. Είναι ένας κύκλος, φαύλο κύκλος. Είναι μια ολόκληρη αλυσίδα που, πάνω στην οποία θα πρέπει να δουλέψουμε. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι νέο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό και το λέτε κι εσείς στην μελέτη σας. Υπογραμμίζετε ότι ήδη το 2011 είναι στη σελίδα 68 της εκθεσή σας. Έλεγε μια μελέτη για στοιχεία και νούμερα στον τομέα της, ε, των μεταφορών. Σε εκείνη την περίφημη αγορά που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση της στόχης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα πορίσματα ήταν πολύ σαφή. Τι έχει γίνει τέσσερα χρόνια μετά? Σας ρωτώ. Τι έχει γίνει κατά τη γνώμη σας. Σήμερα ξαναζητάμε άλλη μελέτη ε, και τα νούμερα είναι προφανή. Αφού αυτά τα στοιχεία τα είχαμε το 2011, πώς τα χρησιμοποίησατε, τα χρησιμοποίησατε ή όχι και πώς γίνεται να επικρατεί μια τέτοια σιωπή απίστευτη για μια μελέτη που τονίζει σημαντικά ζητήματα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη μου ερώτηση αναφέρεται το θέμα των μεταναστών. Θα ήθελα να γνωρίζω αν στους μετανάστες και στους περιοθυροποιημένους πληθυσμούς σημαίνει το ίδιο, γιατί είναι δείκτες που ξέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και για παράδειγμα το θέμα των Ρώμα. Πώς εντάσσεται αυτό το θέμα, αυτό το, αυτό το ζήτημα στη μελέτη σας. Και κάτι ακόμα που είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου, μια τρίτη ερώτηση. είναι, ποια είναι τα επίγοντα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν για να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Διότι ο συνάδελφός σας ανέφερε και άλλο ένα πρόβλημα, είναι το πρόβλημα της δημογραφικής αλλαγής που οδηγεί στο ένα και περισσότεροι πληθυσμοί να μην έχουν πρόσβαση στην κινητικότητα. Ποια μέτρα λοιπόν επιγόντως θα πρέπει να ληφθούν ώστε να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση και υπάρχουν καλές πρακτικές στα αλήθεια. Μπορείτε να μας πείτε σήμερα χώρες ε, όπου λειτουργεί το πράγμα και τι πρέπει να κάνουμε για να ε, διευρύνουμε και να διαδώσουμε αυτές τις καλές πρακτικές. Ευχαριστώ, Πατρίτσια Σουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Είμαι ευτυχής που σήμερα συζητάμε ε, το την ε, κοινωνική ένταξη των δημοσίων, για τις δημόσιες μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για, τα κοινωνικά για τις κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες. Το θέμα αυτό βρίσκω πως δεν έχει συζητηθεί συχνά στο παρελθόν. Συχνά εστιάζουμε στις ε, παραδοσιακές καταστάσεις στην μετακίνηση, ενώ σε τοπικό επίπεδο σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν δημόσιες μεταφορές που είναι προσιτές σε όλους, στους ηλικιωμένους, στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, ε, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Ε, δεν ε, πρόκειται μόνο για την οικονομική πτυχή αυτών των χρηστών, αλλά και για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω την σχέση, τη συσχέτιση μεταξύ δύο πόλεων με δωρεάν δημόσιες ε, μεταφορές, την κορίτσια της ε, Ιταλίας και την κορίτσια της Σλοβενίας, όπου οι δύο τοπικές κοινότητες ε, συνήλθαν σε συμφωνία και ξεκίνησαν αυτή την δωρεάν δημόσια υπηρεσία μεταφορών που χρηματοδοτείται από τους δύο Δήμους. Και αυτό σας το δίνω ως ένα παράδειγμα θα μπορούσε να ακολουθηθεί και αλλού. στην Ευρώπη. Ξεχνά, ξεχνάμε τις ε, περιοχές της Υπέθρου, όπου ο κοινωνικός αποκλεισμός ε, είναι περισσότερο αισθητός και όπου οι κοινωνικές δομές είναι διαφορετικές και ο κόσμος εκεί συχνά έχει προβλήματα στο να, φτάσει στις πόλεις. Δεν υπάρχουν τακτικές γραμμές που συνδέουν με τις πόλεις και δεν υπάρχει ούτε δωρεάν πρόσβαση στις μεταφορές. Στις αστικές περιοχές η κατάσταση είναι διαφορετική. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα αστικά κέντρα και διαφορετική προσέγγιση στις περιοχές της υπαίθρου. Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι πώς θα μπορεί κανείς να μεταβεί από την πόλη στην περιοχή της υπαίθρου εφόσον δεν υπάρχουν ελεφορικές γραμμές για παράδειγμα για άτομα με ειδικέ ανάγκες ή για άτομα από μειονεκτικές ομάδες. Ε, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε καθώς επίσης και το πώς θα παρέχουμε δημόσιες μεταφορές για αυτές τις ομάδες. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι φυσικά σημαντικά. Αυτό το οποίο ωστόσο είναι επίσης σημαντικό είναι να χρησιμοποιηθούν με λογικό τρόπο. Ανέφερα τις τοπικές κοινότητες και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη γι' αυτό. Ευχαριστώ. Λούση Άντερσον. Προτελευταία. Ναι, διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεσή σας. Με ενδιαφέρον διάβασα στη σελίδα 32 ότι οι περισσότερες μελέτες στην Ευρώπη προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Χαίρομαι που έχουμε τόσα δεδομένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. αλλά θεωρώ ότι είναι, έλλειψη, ότι είναι πρόβλημα η έλλειψη στοιχείων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για να έχουμε καλύτερα δεδομένα από όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή ήταν η μία μου παρατήρηση. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε απόψεις όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα σε θέματα μεταφορών, κοινωνικού αποκλεισμού και στέγασης, διότι αυτό είναι θέμα κλειδί. Βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στο, στην κατοικία και στην δουλειά έχουν, έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων και ο κόσμος δεν έχει λεφτά για τέτοιες μετακινήσεις. Η κοινωνική στέγαση λοιπόν ε, όταν αποτελεί επένδυση έχει κοινωνικό αντίκτυπο που σχετίζεται και με τις μεταφορές και όσον αφορά τις τιμές, ε, έχετε έναν πίνακα όσον αφορά την ικανοποίηση με τις τιμές. Αυτό είναι καλό, αλλά τουλάχιστον αν κοιτάξουμε τα στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να αναλύσουμε τα στοιχεία ανάλογα με αυτούς που πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο, για παράδειγμα, ή δεν πληρώνουν καθόλου εισιτήριο. Μπορεί να είναι ικανοποιημένοι επειδή δεν πληρώνουν τίποτα ή επειδή πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν υπάρχουν πιο αναλυτικά στοιχεία ε, ε, στην μελέτη του Ευρωβαρόμετρου όσον αφορά την ικανοποίηση και μιλήσατε για σχετικά επίπεδα. Υπάρχει μια μελέτη και από τα 28 κράτη-μέλη που να συγκρίνει ιδιαίτερα τις αστικές περιοχές ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Εμείς ε, γνωρίζουμε ότι είμαστε από τις χώρες με το πιο υψηλό εισιτήριο λεωφορείων, αλλά μας λένε ότι και στη Μαδρίτη τόσο ακριβά είναι τα ειστήρια. Υπάρχει συγκριτική μελέτη για τις τιμές των εισιτηρίων. Πρέπει να το λάβει κανείς αυτό υπόψη ε, όταν συγκρίνουμε το επίπεδο διαβίωση των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ μία ερώτηση και έχει να κάνει όχι ε, με την δημόσια και ε, ιδιωτική ε, μετακίνηση. Έχει να κάνει και με, με, με μηχανή, έχει να κάνει και ε, με τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Η ποδηλασία δεν στοιχίζει τίποτα. Γνωρίζω πόλεις όπου το 20% των ανθρώπων δεν έχουν χρήματα όχι μόνο για αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουν ούτε και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχετε κάποιο θετικό παράδειγμα ε, σχετικά με το πώς μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ε, να προσφέρουμε εναλλακτική λύση. Πρωτού όμως ε, σας δώσω το λόγο, θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Παρακαλώ. Όχι, η Κομισιόν δεν θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για όλες σας τις ερωτήσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας, διότι μου είπαν ότι έχω στη διάθεσή μου μόνο πέντε λεπτά. Θα ήθελα όμως να πω λίγα πράγματα. Πρόκειται για μια αρχική μελέτη. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να αναλυθούν περισσότερο. Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία που είναι αναλυμένα ανά είδος χρήστη, είδος μεταφορών και άλλα θέματα που αφορούν τα διάφορα είδη χρηστών. Υπάρχουν ε, μελέτες σε πολύ τοπικό επίπεδο, μερικές φορές οι Δήμοι κάνουν έρευνες, έχουμε πολύ λίγα στοιχεία όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα πράγμα που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να βελτιώσουμε την συλλογή στατιστικών στοιχείων, να βελτιώσουμε την ποιότητα των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα βασικά προβλήματα όταν μιλάμε για μεταφορές και κοινωνική ένταξη. Υπάρχει και ένα θέμα που συνδέεται με την έρευνα. Αυτή τη στιγμή οι νέες τεχνολογίες δεν μπορούν να ε, αλλάξουν ε, την κατάσταση, αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα. Έχουμε το πρόγραμμα Horizon 2020, για παράδειγμα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην έρευνα νέων τεχνολογιών που προωθούν την κοινωνική ένταξη. Και εδώ υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό θέμα που θύχτηκε στη συζήτηση κατά την εξέταση των μελετών αντικτύπου των διαφόρων πολιτικών. Κάθε φορά που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προτείνουν μια νέα πολιτική πρέπει να εκπονήσουν και μελέτη αντικτύπου. Σε αυτές λοιπόν τις μελέτες αντικτύπου θα πρέπει να εξετάζουμε όχι μόνο το βραχυπρόθεσμο κόστος και όφελος, το οικονομικό, θα πρέπει όμως να εξετάσουμε και τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές συνέπειες πέρα από τις περιβαλλοντικές. Εάν δεν εξετάσουμε τις κοινωνικές συνέπειες, τον κοινωνικό αντίκτυπο, υποτιμούμε το ενδεχόμενο κόστος κάποιων επιλογών όταν καθορίζουμε τις πολιτικές μεταφορών. Εάν εξετάσουμε μόνο την βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και οικονομική βιωσιμότητα, αυτό σημαίνει ότι δεν εξετάζουμε τους κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού που μπορούν να επιφέρουν υψηλότερο κόστος στο μέλλον, διότι στο τέλος θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να πεθάνουν, ούτε θα εξαφανιστούν από μόνοι τους. Όταν λοιπόν εξετάζουμε τον, αντίκτυπο διαφόρων πολιτικών και ιδιαίτερε πολιτικές μεταφορών όπου συνήθως δεν εξετάζουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο στις μεταφορές, στις υποδομές, θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ περισσότερο τον κοινωνικό αντίκτυπο σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Η ανάλυση κόστους όφελους θα πρέπει να εξετάσει λοιπόν και το κοινωνικό όφελος και κόστος, όχι μόνο το οικονομικό. Άλλο θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μία απάντηση που να καλύπτει όλους. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες στην κινητικότητα. Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας μπορεί να ανταποκρίνεται σε κάποιες ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρίες, τους ηλικιωμένους κλπ. Δεν μπορεί όμως να καλύψει όλες τις ανάγκες τους. Υπάρχουν κάποια πιλωτικά προγράμματα πληροφόρησης από πλευράς ε, των αρχών που είναι αρμόδιες για τις μεταφορές για να παρέχονται πληροφορίες σε τυφλούς, για παράδειγμα, ή άτομα με άλλες αναπηρίες. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τον ρόλο των τοπικών αρχών. Τα περισσότερα από τα προγράμματα που περιγράφονται στο έγγραφο εφαρμόζονται από τις τοπικές αρχές, διότι αυτές μπορούν καλύτερα να διαπιστώσουν ποιες είναι οι ανάγκες και να ανταποκριθούν σε αυτές. Το πρόβλημα είναι ότι κατά τις περικοπές του προϋπολογισμού οι πρώτοι που πλήττονται είναι οι τοπικές αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό όσον αφορά τη δημογραφική αλλαγή και τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Θα αυξηθούν αυτές οι τάσεις στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να τις αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης, οι χώρες που ασχολούνται ε, πιο λίγο καιρό με το πρόβλημα αυτό όπως είναι η Ιταλία, μπορούν να μάθουν από τις χώρες ε, που έχουν περισσότερη εμπειρία, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, όπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερη παράδοση μετανάστευσης και μπορούμε να μάθουμε και από τις αρνητικές εμπειρίες τους ε, για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Νομίζω ότι οι, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να, να κάνουν πολλά στον τομέα αυτόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μετανάστευσης θα μπορούσαν να παίξουν πολύ πιο ε, έντονο ρόλο συντονισμού κατά την ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών. Θα μπορούσαν επίσης να εκπονήσουν κάποια πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά για παράδειγμα την προσβασιμότητα, την ασφάλεια. Και θα μπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν τους πολιτικούς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο απέναντι στα θέματα κοινωνικής ένταξης όταν καθορίζουν τις πολιτικές αυτές. Για παράδειγμα, με την ανταλλαγή των πρακτικών, με βελτίωση της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της συλλογής δεδομένων. Μπορούν να προωθήσουν την καλύτερη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Μπορούν δηλαδή να λένε ότι θα πρέπει να εξετάζει κανείς ε, το θέμα αυτό κατά την χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Πολλές προτάσεις λοιπόν ε, μπορεί να υποβάλει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο προς ε, την Κομισιόν, προς τα κράτη-μέλη και προς όλους τους παράγοντες των τομέα αυτών. Λυπάμαι που δεν πρόλαβα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και για την μελέτη και για την παρουσίαση που μας κάνατε. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε πολλή δουλειά λοιπόν για να εφαρμοστούν όλα αυτά στα προγράμματα των κρατών μελών και της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ θερμά. So, έτσι στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το πακέτο της Ενεργειακής Ένωσης. Πρωτόκολλο του Παρισιού. Και δίνω πρώτα το λόγο στους εισηγητές και πρώτα οι κυρίες, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόκειται για τη γνωμοδότησή μας για την Ενεργειακή Ένωση. Η ε, αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η ΙΤΡΕ στο Κοινοβούλιο και η ΙΤΡΕ έκανε τη συζήτηση της ε, σήμερα το πρωί για την έκθεση αυτή. Θα πρέπει να σας πω ότι ο τομέας των μεταφορών δεν περιλαμβάνεται ακόμα στη σχέδια έκθεσης, οπότε θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ώστε να συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση. Θα πρέπει να σας πω ότι για την Ενεργειακή Ένωση ο τομέας των μεταφορών είναι πολύ σημαντικός γιατί αντικατοπτρίζει πάνω από το 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Πάνω από το 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στον τομέα των μεταφορών. Και είναι αυτός ένας στόχος αν θέλουμε να έχουμε ασφαλή και βιώσιμη αλλά και προσιτή ενέργεια για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο τομέας των μεταφορών όμως βασίζεται περισσότερο ε, κατά 94% στα προϊόντα πετρελαίου για την ενέργεια που καταναλώνει. Έχουμε πολλά να κάνουμε λοιπόν. Πρέπει να βρούμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ω προς το κόστος για να περιορίσουμε τις εκπομπές και είναι ιδιαίτερα αυτό σημαντικό στις αστικές περιοχές όπου ζουν το 70%, ζει το 70% των ευρωπαϊκών λαών. Όπως ε, είπαμε και νωρίτερα, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε για το σχεδιασμό των πόλεων. Σύντομα θα σας αναφέρω αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί είναι μια γνωμοδότηση, δηλαδή πρέπει να είναι πολύ σύντομη. Μπορούμε να υπογραμμίσουμε μόνο κάποια σημεία, πρέπει να είναι μικρότερη από μια σελίδα η τελική μας γνωμοδότηση. Οπότε μπορούμε απλά να τερνώσουμε άλλα, ε, κάποια μόνο στοιχεία. η αποδοτικότητα και επάρκεια στην ενέργεια είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους του πακέτου για την ενέργεια και η ιδέα μετακίνησης προς τους πιο αποτελεσματικούς, μάλλον αποδοτικούς ε, τρόπους μεταφορών όπως οι σιδηρόδρομοι, οι εσωτερικές πλωτές οδοί ε, είναι πολύ σημαντική αλλά όπως ξέρουμε αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε και τις οδικές μεταφορές στο μέλλον αλλά και τέτοιου είδους οδικές μεταφορές που να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον από ό,τι σήμερα. Πιστεύω πως έχουμε καλές δυνατότητες για να το πετύχουμε αυτό. Ε, εξαρτώμεθα πολύ από το πετρέλαιο ακόμα στον τομέα των μεταφορών, αλλά ήδη έχουμε διάφορες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες και πολλά καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον. Ο ταχύτερος τρόπος λοιπόν για να περιοριστούν οι εκπομπές είναι αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα από τα ανανεώσιμα καύσιμα, την τον ηλεκτρισμό από άλλες εναλλακτικέ χαμηλής εκπομπής ε, άνθρακα. Θα πρέπει να γίνουν ε, ε, επενδύσεις στην έρευνα, στην παραγωγή και στη διανομή των ανανεώσιμων καυσίμων. καθώς επίσης και στις σύγχρονες τεχνολογίες. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια για την απανθρακοποίηση του τομέα των μεταφορών. και να μείνουμε μπροστά πάντα από τους, από τους ανταγωνιστές μας. Ένας τρόπος ε, θα ήταν ίσως να ανοίξουμε την αγορά ε, και της αεροπλοείας ε, ή της ναυσιπλοείας είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι είναι παγκοσμιοποιημένοι τομεί και άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε κανόνες ε, διεθνώς στη Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας ώστε να ε, θεσπιστούν ε, κοινοί στόχοι για την μείωση των εκπομπών σε σχέση με την αυσιπλοεία, η στήριξη για την έγκαιρη ανάπτυξη του υγροποιημένου φυσικού αερίου χρειάζεται στην Ευρώπη. Και πρόεδρε, συνάδελφοι, ψηφιοποίηση δεν θα πρέπει να την ξεχνάμε όταν μιλάμε για ενεργειακή επάρκεια στην Ευρώπη. Ε, αυτές οι νέες τεχνολογίες και τη ψηφιοποίηση δίνουν νέες ευκαιρίες για νέες ευφυείς υπηρεσίες μεταφορών. Θα πρέπει αυτά να ληφθούν υπόψη, αυτή η πτυχή μάλλον να ληφθεί υπόψη, καθώς και να εστιάσουμε στις δυνατότητες που προσφέρει αυτός ο τομέας. Όπως γνωρίζουμε, η ευφυείς και η κυκλοφορία είναι επίσης πιο αποδοτική ως προς την ενέργεια, τη χρήση της ενέργειας. Οι ομαλές υποδομές για την κυκλοφορία είναι πολύ σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αλλά και για την αποδοτική εσωτερική αγορά. Πάντοτε θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους προώθησης της ε, ε, των καθαρότερων τρόπων μεταφοράς, δημιουργώντας και θέσεις απασχόλησης για τους Ευρωπαίους. Οπότε, Πρόεδρε, εδώ έχω τα βασικά σημεία που θέλω να τονίσω ε, ε, για τον τομέα των μεταφορών ως τμήμα της Ενεργειακής Ένωσης, αλλά ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος για την δική μας Επιτροπή είναι να θυμίσουμε και να υπογραμμίσουμε πόσο μεγάλο τμήμα ε, ε, της Ενεργειακής Ένωσης είναι ο τομέας των μεταφορών, ότι πρέπει δηλαδή να προσεχθεί ιδιαίτερα και να κινηθούν οι επενδυτές όλου αυτού του τομέα σε χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να ευχαριστήσω τώρα όλους τους και ηγητές. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ε, για τη συνεργασία και προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση και στις παρατηρήσεις σας για αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι ο δεύτερος κλάδος του ενεργειακού πακέτου που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια ανακοίνωση εν ώψη του Παρισιού όπου θα λάβει η χώρα η 21η διάσκεψη των μερών για το κλίμα στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Υποτίθεται ότι θα ήταν η διάσκεψη η οποία θα κατέληγε σε συμφωνία το 2015, μια ελπίδα που έχουμε από την Κοπενχάγη και το 2009. Θεωρείται ότι έξι χρόνια μετά θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια διεθνή συμφωνία όπου από το, 20, το 2020 και πέρα όλες οι χώρες θα εμπλακούν στον αγώνα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ανθρώπινας δραστηριότητα στο κλίμα. Βεβαίως η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει το φάκελο, αλλά και εμείς πρέπει να δούμε το θέμα από τη σκοπιά των μεταφορών. Πρέπει να έχουμε την έκθεση της σχετικής Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Ε, έχω την εντύπωση ότι ο τομέας των μεταφορών δεν είναι εξαιρετικά διαθέσιμος. Αν μιλούμε για διαφορετικούς ε, τομείς, τότε συχνά ξεχνούμε τον τομέα των μεταφορών και για το κλίμα. Είναι περίεργο να τα ξεχνούμε κάτι τέτοιο, γιατί αν δούμε τους ευρωπαϊκούς στόχους και ε, αν εντοπίσουμε επιτυχίες σε όλους τους τομείς οικονομίας, δηλαδή ε, οι μεταφορές είναι οι μόνες που συνεχώς οι εκπομπές τους αυξάνουν τα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ όλοι οι άλλοι κλάδοι της ε, ε, θερμοκρασίας. Ε, όλοι οι άλλοι κλάδοι της οικονομίας, με συγχωρείτε, απομακρύνονται από τον άνθρακα και μειώνουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Και είναι ένα μήνυμα, μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, αυτό που πρέπει να σταλεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο Παρίσι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διεθνή αεροπορία και στη διεθνή ναυτιλία. Ξέρουμε όλα αυτά που έχουν προαναφερθεί. Έχουμε δύο διεθνείς οργανώσεις, φορείς που είναι υπεύθυνοι, είναι αρμόδιοι. Η, η ΚΑΟ για την αεροπορία, η IMO, η ΙΜΟ για την αυτιλία. Και τα λέω, ξέρετε, με πολύ εύηχο τρόπο. Θα έπρεπε να μιλήσω πολύ πιο κατηγορηματικά. Να σας πω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος έστειλε μια αντιπροσωπεία στον ΙΜΟ, στον IMO, πριν από δύο εβδομάδες στο Λονδίνο, όπου συζητήθηκαν τα δεδομένα της διεθνούς ναυτιλίας, αλλά και έγινε και συζήτηση αν θα πρέπει να τεθεί στόχος για τη μείωση των αερίων φαινομένου θερμοκηπίου. Έγινε συζήτηση εντός του IMO. Ήταν, ήταν μια πρόταση από τις νήσους Μάρσαλ, ε, μια χώρα που έχει πάρα πολλά πλοία, έχει πάρα πολλούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας. Όμως, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας θέλουν να προλάβουν το πρόβλημα, γιατί ε, είναι η περιοχή που έχει χτυπηθεί από την κλιματική αλλαγή. Ξεκινάει λοιπόν η συζήτηση για το κλίμα και στο εσωτερικό του IMO, και την επόμενη χρονιά η ΚΑΟ, η Διεθνής, ε, ο Διεθνής Οργανισμός για τη Διεθνή Αεροπορία, θα πρέπει τουλάχιστον να δημοσιεύσει ένα σχέδιο για τη μείωση τέτοιου είδους εκπομπών. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αν πάμε προς μια ειδική γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών για ε, την ανάγκη ανάληψης διεθνούς δράσης για τα θέματα του κλίματος ή γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ε, τουλάχιστον εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών πρέπει σίγουρα να έχουμε εξετάσει το πώς ο IMO και ο ICAO θα συμβάλλουν για να μην αυξηθεί η παγκόσμια θερμοκρασία κατά δύο βαθμούς ή να μειωθεί κιόλα. Ε, βεβαίως με τις τροπολογίες μπορούμε να επιδείξουμε ευελιξία για να δούμε τι θα δούμε. Όμως νομίζω ότι η γνωμοδότηση αυτή παρουσιάζει τα πιο σημαντικά θέματα, το θέμα της τιμολόγησης, το θέμα του, της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, της ε, ε, απελευθέρωσης από τον άνθρακα και τα ορυκτά καύσιμα ότι δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, έχει να κάνει και με τα logistics, την επιμελητία, τον εφοδιασμό και την ηλεκτροποίηση, τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών. Το σημαντικό είναι οι τιμές να είναι σωστές και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο διεθνές στερέωμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την περασμένη εβδομάδα ε, έδωσε ένα νούμερο. Οι επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα όχι μόνο στο τομέα των μεταφορών αλλά παντού, συνολικά στον κόσμο ετησίως δίνουμε 5.300 δολάρια επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων ε, και αυτό παραμένει τεράστιο πρόβλημα εάν θέλουμε να κάνουμε τη μετάβαση προς μια οικονομία που θα εξαρτάται όλο και λιγότερο από τον άνθρακα. Στην έκθεση, στη γνωμοδότηση προβάλλω αυτό το επιχείρημα, αλλά θα το αναπτύξουμε έτσι περαιτέρω όταν δεχθούμε τις τροπολογίες οι οποίες μπορούν να κατατεθούν μέχρι και τις 5 Ιουνίου. Ανυπομονώ να έχουμε την ε, συμβολή των συναδέλφων να έχουμε μια σωστή γνωμοδότηση με την οποία να τροφοδοτήσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος η οποία ασχολείται με τη διάσκεψη των μερών του ΟΗΕ την 21η στο Παρίσι. Και έτσι ο, ο κλάδος των μεταφορών θα τύχει της προσοχής που του αξίζει. Η Κριστίν παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω για την εξονόματο στη Τερέζα για την Ένωση την Ενεργειακή ε, που δυστυχώς ε, έλειπε, ε, λείπει γιατί είχε κάποια άλλη ενελειμμένη υποχρέωση. Καταρχήν λοιπόν θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την εργασία της και για το ευχαριστίες που έδωσε στους, μάλλον και για τη συνεργασία με τους Κιώδης. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική, θα αλλάξει το ενεργειακό περιβάλλον στα επόμενα χρόνια. Ορίζοντα που προετοιμάζουμε θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ε, στην ε, Ένωση. Ελπίζουμε πως η Επιτροπή Ήτρε θα λάβει υπόψη αυτήν την ε, έκθεση Η Τερέζα Γκρίφιν θεωρεί πως οι απόψεις της κυρίας Φεργίνου για την ενίσχυση της ηλεκτρικής ε, κινητικότητας και η ηλεκτροδότηση των ε, μέσων μαζικής μεταφοράς κινούνται προς σωστή κατεύθυνση. Η Ένωση Ενεργειακή θα πρέπει να πλαισιώνεται από ένα σύστημα οριζόντιας διακυβέρνησης, το οποίο είναι σταθερό και διαφανές. Αυτό το σύστημα θα πρέπει επίσης να τον προωθεί το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτών και των τοπικών αρχών. Ε, ε, εδώ ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει προσβασιμότητα σε όλα τα είδη μεταφορών. Να προωθηθούν επίσης δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τις υποδομές που ευνοούν ε, τους βιώσιμους ε, τρόπους μεταφορών. Η Τέρεζα Γκρίφιν ε, μπορεί να συνεργαστεί μαζί σε τη συνέχεια αυτής της έκθεσης και είναι βέβαιη ότι μια ισορροπημένη γνωμοδότηση θα συνταχθεί τελικά. Και τώρα περνώ στο πρωτόκολλο των Παρισίων. Για την COP21 πρόκειται για ένα έγγραφο αναφοράς ε, με το οποίο θα πρέπει να συμμορφωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην COP21. Θα πρέπει να είμαστε απαιτητικοί και να στείλουμε συγκεκριμένο μήνυμα στη Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελήσει την αιχμή του δόρατος για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτάσει να περιληφθεί στο πρωτόκολλο των Παρισίων στόχοι που να είναι δεσμευτικοί για να περιοριστεί η θέρμανση του πλανήτη στους δύο βαθμούς και να μειωθούν οι εκπομπέ του διοξιδίου του μάλλον αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% μέχρι το 2050 ε, ε, σε σχέση με τις εκπομπέ του 2010 είμαστε σύμφωνοι. Μείωση επίσης των εκπομπών ε, από τον τομέα των μεταφορών. Όπως υπόθηκε, Ε, εδώ ε, πρέπει να τα πούμε όλα σύντομα και γρήγορα γιατί ε, υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος της νομοδότησης. Θα πρέπει να τονιστεί η ιδιαιτερότητα των μεταφορών όχι μόνο στον κορμό του πρωτοκόλλου αλλά και στις παράλληλες πρωτοβουλίες όπως η ατζέντα της COP21 με καινοτόμες και συγκεκριμένες λύσεις. Σε αυτή την προοπτική θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η χρηματοδότηση και τα μέσα που θα δημιουργηθούν για να χρηματοδοτηθούν οι κλιματικέ πολιτικέ, θα πρέπει να δώσουν τα κονδύλια προ τον τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, επειδή πάνω από το 70% του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές και οι εκπομπέ σε αυτές τι περιοχές αντιπροσωπεύουν το 1 τέταρτο των εκπομπών του τομέα των μεταφορών, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τα διακυβεύματα της, ε, κινητικότητα, της βιώσιμης ε, κινητικότητας στα αστικά κέντρα μέσα στην ατζέντα τη COP21. Οι δε που θα προβλεφθούν δεν θα πρέπει να περιοριστούν μόνο στην ηλεκτροδότηση των τρόπων μεταφορών, αλλά να σκεφτούμε και άλλο είδου οχήματα, όπως αυτά που ε, κινούνται με φυσικό αέριο ή με βιοαέριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα και ω εκ τούτου θα πρέπει αυτό Αυτές οι ε, πρωτοβουλίες που θα προκύψουν από το πακέτο Ενέργεια 2030 και ιδιαίτερα για τις οδικές μεταφορές θα πρέπει να στοχεύουν στην σημαντική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για τα βαριά και ελαφρά οχήματα ώστε να μειωθούν κατά 20 με 30% οι σχετικές εκπομπές μέχρι το 2030. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ιβο Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι εισηγητής της Επιτροπής ΕΝΒΗ για την Ενεργειακή Ένωση. Θα μιλήσω εδώ όμως ως σκιώδης εισηγητής για το πρωτόκολλο του Παρισιού. Καταρχάς θα πω ότι η πολιτική μας ομάδα συμμερίζεται πολλές από τις ανησυχίες που εξέφρασε ο εισηγητής στη γνωμοδότησή του, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενίσχυση των ηλεκτροκίνητων μέσων και την επιτάχυνση προς τον σκοπό αυτόν. Θα ήθελα, όπως είπε ήδη ο εισηγητής και γι' αυτό μπορώ να είμαι πολύ σύντομος, θα ήθελα να επικεντρωθώ στην αεροπλοεία Πρέπει εδώ να γίνουν πολλές δεσμεύσεις από διάφορες πλευρές, αλλά υπάρχει πλήρης έλλειψη προόδου στους οργανισμούς αυτούς. Θα πρέπει να πετύχουμε κάποια πρόοδο πριν το τέλος της επόμενης χρονιάς, το οποίο όμως θα έρθει πολύ σύντομα. Η πρόοδος λοιπόν των διεθνών οργανισμών στο θέμα αυτό ήταν πάρα, πάρα πολύ αργή. Όσον αφορά το πρωτόκολλο του Παρισιού θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι είναι απαραίτητες οι δεσμεύσεις από τους διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη την αργή έως και μηδενική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα. Θα ήθελα στον και του συναδέρφους να πω ε, επίσης ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ευαίσθητο θέμα της φορολογίας ε, του τομέα της αεροπλοΐας. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα προνόμια του τομέα αυτού, διότι μιλάμε για ΦΠΑ και φόρο στα καύσιμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τομέας αυτός χαίρει προνομιακής αντιμετώπισης. Η μείωση αυτών των παρεκκλήσεων ε, θα σημάνουν συνθήκες ίσου ανταγωνισμού σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφορών. Και έτσι θα δημιουργήσουμε και μια δυνατότητα μεταφοράς ε, των φόρων. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό, αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα των εναλλακτικών καυσίμων. Ήδη αναφέρθηκε η υποδομή για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Θα υπάρξει βέβαια μια επικάλυψη ανάμεσα στην έκθεσή σας και την Λευκή Βίβλο. Ευχαριστώ πολύ, Κοσμοσοτόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συγητή για την γνωμοδότηση αυτή. Στον τομέα της κλιματικής πολιτικής οι μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο, γι' αυτό είναι σημαντικό το ότι μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε στο θέμα αυτό. Οι μεταφορές είναι ο μόνος τομέας όπου αυξάνονται οι εκπομπές και έτσι χειροτερεύουν οι στατιστικές. Όλοι οι πολίτες χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς και όλοι συμβάλλουν στην αύξηση των εκπομπών. Έχουμε τους φιλόδοξους στόχους του πρωτοκόλου του Παρισιού. Τα ορυκτά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών αποτελούν πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε το περιβάλλον, αλλά οι τιμές αυτών των καυσίμων είναι καλές. Αυτό σχετίζεται με όλους τους τρόπους μεταφορών. Όλοι αναζητούν εναλλακτικά καύσιμα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να επιβαρυνθούν υπερβολικά στο θέμα αυτό. Κατά την εξέταση των αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να ληφθούν διάφοροι παράγοντες υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ομοιόμορφη. Οι συνθήκες διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Οι τιμές των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Πολωνία θα αυξηθούν ε, πολύ περισσότερο αν χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικέ μορφέ ενέργεια, ε, διότι ε, το 90% τη ενέργεια παράγονται από το λιγνίτη. Στη Σουηδία θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε με τέτοιο κόστο τι οικονομικά στενέστερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε το κόστος των υποδομών και την πρόσβαση στις πιο απόμακρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να κατασκευάσουμε δρόμους, ε, σιδηρόδρομους, θέλουμε πιο γρήγορες μεταφορές. Είναι σημαντικά όλα αυτά, αλλά τον στόχο της, ο στόχος της μείωσης ε, των εκπομπών δεν επιτρέπεται να εμποδίσει την πραγματοποίηση προγραμμάτων κλειδιά, όπως είναι οι άξονες που θα συνδέσουν ε, την Ανατολική με τη Δυτική Ευρώπη. Τρίτον, οι υπηρεσίες στον χώρο των μεταφορών θα πρέπει να προστατεύονται, θα πρέπει να έχουμε ευφυείς λύσεις. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, το καμποτάζ. Θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις υπάρχουσες δυνατότητες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο των μεταφορών ε, στο ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ, Νασιοφάρια. <clears throat> Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την γνωμοδότηση ε, και για την, ε, το πνεύμα συνεργασίας που έδειξε από την αρχή της διαδικασίας. 94% ε, εξαρτάται ο τομέας των μεταφορών από τα, από τα ορυκτά καύσιμα. Το θέμα της ε, απαλλαγής από τον άνθρακα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής κατά των κλιματικών αλλαγών. Μια τέτοια προσέγγιση έχει θετικές, ε, ε, θετικά πλεονεκτήματα, όχι μόνο σε σχέση με την κλιματική πολιτική, αλλά και για να βελτιωθεί η ενεργειακή επάρκεια για τις μεταφορές και να μειωθεί η εξωτερική εξάρτηση για την, ε, από, ε, για την ενέργεια. Θα πρέπει να προωθηθούν οι επενδύσεις στις νέες πιο καθαρές τεχνολογίες μεταφορών και να γίνουν επενδύσεις στις τεχνολογικές έρευνες. Βέβαια, οι νέες τεχνολογίες είναι ένα από τους σημαντικούς τομείς από τη στιγμή που μπορούν να ενσωματώσουν μορφές ανανεώσιμες ενέργειες και που θα μπορέσουν έτσι να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στη αστικά κέντρα, μειώνοντας το θόρυβο και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα. Η προώθηση των, τεχνολογιών, των καθαρών τεχνολογιών θα είναι ευνοϊκή και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ώστε να μείνει στην πρωτοπορία τη τομέα αυτού. Η διαδικασία τυποποίησης αλλά και της ε, χρηματοδότησης θα επιτρέψει στις καινοτόμες ε, ε, εταιρείες να εκμεταλλευτούν την ενιαία αγορά. Επίσης θα μπορέσει έτσι να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό των συλλογικών μέσων μεταφοράς γιατί ε, ακριβώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν συστήματα εναλλακτικά για τη λειτουργία τους, αλλά και να χρησιμοποιήσουν ευφυή e e συστήματα ψηφιακά ε, για να μπορέσουν να ε, είναι πιο αποδοτικά και να παρέχουν στους πολίτες πιο ελκυστική υπηρεσία. Συμφωνώ δε και με την εισηγήτρια όσον αφορά την ανάγκη εθάρρυνσης σε πιο αποτελεσματικών, πιο αποδοτικών μέσων μεταφορών, όπως οι σιδηρόδρομοι ή οι ε, εσωτερικές πλωτές οδοί ή η ναυσιπλοεία. Χρειάζονται επενδύσεις στα λιμάνια μας, καθώς και στα σιδηροδρομικά μας δίκτυα, ώστε να γίνει η μετακίνηση ε, των μεταφορών προς αυτά τα είδη μεταφορών. Τώρα, όσον αφορά την μετάβαση, το φυσικό αέριο, στηρίζω την ε, ένταξή τους στην ε, διαδικασία και στις συνθήκες ε, που θέλουν να βελτιώσουν τη γεωστρατηγική μας θέση σε σχέση με άλλες περιοχές. Πάντως, δεν θα πρέπει να θα πρέπει μάλλον να προωθηθεί η χρήση του φυσικού αερίου στις, μεταφορές, στις δημόσιες μεταφορές. Έχω εδώ μια διαφωνία τώρα σε σχέση με αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί δεν υπάρχουν αρκετές ε, φιλοδοξίες όσον αφορά τη μικρότερη χρήση ε, διοξιδίου του άνθρακα, εκπομπή μάλλον διοξιδίου του άνθρακα από την αεροπλοεία και την αυσιπλοεία. Ενώ ε, γίνεται προσπάθεια για να φτάσουμε σε μια διεθνή συμφωνία όσον αφορά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου για για την αυσιπλοεία. Μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδο. θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Ναύση Πλοίας ε, οι προτάσεις που έγιναν έχουν ε, απορριφθεί. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξουμε, να, μάλλον, να επιμείνουμε για δημοκρατικές διαδικασίες. Θα πρέπει να αναλυφθεί μια διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε αλλαγές και προόδους στη Διεθνή Οργανισμό Ναυσιλίας, να αναλάβει την πρωτοβουλία η Ένωση για τον εξυγχρονισμό των εκπομπών του Ισναυσιπλίου σε ένα πρώτο ε, μικρό βήμα ο ορισμός προθεσμιών και στόχων είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το τομέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει το κύριο της για να προχωρήσουν τα πράγματα. Τώρα, δύο λόγια για τις επενδύσεις. Χρειάζονται επενδύσεις που θα στηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων και θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία και πόλη πιο ε, βιώσιμες, ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και από εναλλακτικές πηγές. Σε σχέση με την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και άλλες πηγές χρηματοδότησης, θα πρέπει να ε, προτιμήσουμε τη χρηματοδότηση για τις σιδηροδρόμους, τις ε, θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και τις εσωτερικές πλωτές οδούς, καθώς και τις επενδύσεις στα λιμάνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά και την εισηγήτρια και να της πω ότι είμαστε ως στη διάθεσή της για να τα συζητήσουμε ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την τελευταία στιγμή μου ζητήθηκε να μιλήσω εξ ονόματος της κυρίας Γκεζίνα Μάισνερ δεν το περίμενα το πρωί. Είχα άλλες υποχρεώσεις. Επομένως δεν θα κάνω προσωπικά σχόλια. Θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω κάποιες τροπολογίες που υποβάλλει στον εισηγητή. Και θα ήθελα να διαβάσω τα, τις παρατηρήσεις της Γκεζίνα. Θέλουμε και ευχόμαστε στο Παρίσι να εξευρεθεί μια νομικός δεσμευτική συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι προφανές ότι η φιλοδοξία και η ανησυχία για το Παρίσι είναι κάτι το οποίο όλοι βιώνουμε. Ελπίζει η Κεζίνα ότι όσο πιο πολλοί εταίροι ε, συμπράξουν και συμπορευτούν, τόσο καλύτερη θα είναι η συμφωνία. Ο κλάδος των μεταφορών είναι πηγή εκπομπών αερίου φαινομένου θερμοκηπίου. Ορισμένοι κλάδοι του, υπόκλάδοι των μεταφορών έχουν καταβάλει πολλή προσπάθεια, κάποιοι άλλοι πολύ λιγότεροι. Η Ευρώπη δεν πρέπει να προχωράμε μονομερείς υποχρεώσεις από τη στιγμή που δεν υπάρχει παγκόσμια συμφωνία. Αν εμείς στηρούμε μονομερείς υποχρεώσεις, αυτό θα είναι τεράστιος κόστος ε, για την ευρωπαϊκή οικονομία χωρίς να έχουμε συγκρίσιμα ωφέλη για το κλίμα. Ε, ξέρουμε από παρελθούσα εμπειρία ότι τα μονομερή μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά. Ας μην επαναλάβουμε το λάθος που έχουμε ήδη διαπράξει σε άλλους τομείς. Και αναφέρεται και η Ζήνα στο τομέα της ναυτιλίας. Όσο περισσότερα κράτη προσχωρήσουν στη συμφωνία τόσο λιγότεροι είναι οι κίνδυνοι. Αυτά λοιπόν είναι τα σχόλια της Γκεζίνα. Ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας και σε ό,τι με αφορά θα υποβάλω τις δικές μου τροπολογίες μαζί με τους άλλους συναδέλφους σε εύθετο χρόνο. Η Μαρία Κίλουγκ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χάρη και στους δύο εισηγητές πολλές τροπολογίες υποβάλλουμε και θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή των δύο εισηγητών. Καταρχάς η Ενεργειακή Ένωση συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος της παραγωγής ενέργειας πρέπει να τύχει μεγαλύτερης και περισσότερης προσοχής εδώ. Θα πρέπει να τονιστούν περισσότερο οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας που μπορούν να διαδραματίσουν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Ε, είναι το θέμα τι ενεργειακό μείγμα χρησιμοποιούμε. Πιστεύω ότι οι έξυπνες μεταφορές της πόλης είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και λόγω του όγκου των χρηστών. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε στην Ευρώπη μεταφορές που να χρησιμοποιούν με λογικό τρόπο τον διαθέσιμο χώρο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και κάτε με όλες οι υπηρεσίες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους την ανάγκη οι εκπομπές να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Ας αναζητήσουμε τις λύσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, θα μας στείλετε ε, φιλικές επιστολές μας λέτε το ότι αυτές ε, θα δημοσιεύονται, δεν το περίμενα. Ο Πίτερ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι... Είχα ακούσει τα πάντα στην Επιτροπή μας όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Λε, σήμερα ακούω κάποιον που λέει ότι με απορρίθμιση θα έχουμε μεγάλα κέρδη αν πέσουν οι μεταφορές στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Είστε τυφλός απέναντι στο, στα όσα συμβαίνουν ε, στην ε, πραγματικότητα. Βλέπουμε ανθρώπους με πολύ χαμηλό μισθό και λέτε ότι πρέπει να απορριθμίσουμε ακόμα περισσότερο τώρα τις ε, αγορές μεταφορών. Στη Σουηδία προσέχουμε το περιβάλλον, χρησιμοποιούμε δίζελ στην Σουηδία, στα φορτηγά, από ανθρώπους που εργάζονται υπό συνθήκες σκλαβιάς, δεν έχουν καλά, καλά ε, χρήματα για να φάνε και Ακούω σήμερα ότι με απορρίθμιση των αγορών θα ε, έχουμε μόνο κέρδη. Αξιοπρέπεια δεν έχετε. Οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Μην έρχεστε να μου πείτε εγώ που εργάζομαι 30 χρόνια στον τομέα αυτόν λέγοντας μου ότι με την απορρίθμιση θα κερδίσουμε. Ανικανότητα από πλευρά σας είναι να λέτε τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχει όμως ο καθένας σε δικαίωμα στην ελευθερία λόγου. Η Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει αυτή τη γνωμοδότηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η Ενεργειακή Ένωση ως ιδέα, ως κόνσεπτ είναι κάτι το πολύ περιεκτικό, πολύ ολοκληρωμένο. Είναι διάστατο, είναι ένα έργο που ξεπερνά την ενέργεια, περιλαμβάνει και το κλίμα και τη Γενική ε, Διεύθυνση για τις Αγορές και τη Γενική ε, Διεύθυνση για την Έρευνα και την Τεχνολογία και Καινοτομία περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Έχουμε αρκετές δράσεις, 43 δράσεις ήδη έχουμε προτείνει και ήδη 7 προτείνουμε να γίνουν το 2016 στον τομέα των μεταφορών. Από πλευράς λοιπόν Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφές ότι οι μεταφορές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, είτε πρόκειται για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου κατά 40% σίγουρα πρέπει να ε, ε, ενθαρρύνουμε το πακέτο των μεταφορών και να ενθαρρύνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καλωσορίζουμε τη συμβολή της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να είναι προϊόν διαλόγου με το Κοινοβούλιο και με τους πολίτες. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερο η στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε καταστήσει σαφές εξ αρχής ότι η νέα διακυβερνητική δομή θα πρέπει να είναι σε στενή συνεργασία με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών για να υπάρξει ένας ευρύτερος διάλογος για την ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διαχείρισης και διακυβέρνησης, ένα νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών για να επιτύχουμε τους διαφορετικούς τους διαφόρους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης με την καθοριστική συμβολή του τομέα των μεταφορών. Τώρα, για την γνωμοδότησή σας ε, συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό με την άποψη του εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ελίνα Βάτραμα, από την Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα. Thank you, Mr. and... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα στους Ευρωβουλευτές. Η Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα θέλει να σας ευχαριστήσει για τη γνωμοδότηση. Επικροτεί τη γνωμοδότησή σας και σας ευχαριστούμε και για τις σημερινές σας παρεμβάσεις που δείχνουν το βάθος και το εύρος της κατανόησής σας των σχετικών θεμάτων. Η ανακοίνωση για το πρωτόκολλο του Παρισιού αποτελεί σημαντικό στοιχείο του πακέτου για την Ενεργειακή Ένωση που υιοθετήθηκε από το Σώμα των Επιτρόπων στις 26 Φεβρουαρίου. Έχουμε λοιπόν κάτι εδώ πέρα το οποίο ταιριάζει απόλυτα με την Ενεργειακή Ένωση. Το, το πρωτόκολλο του Παρισιού περιλαμβάνει και ένα όραμα για την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας. Περιλαμβάνει όλους τους τομείς της οικονομίας. Θέλουμε δράση σε όλους τους τομείς της οικονομίας, σε όλες τις μεγάλες οικονομίες και θέλουμε να σεβαστούν τους όρους της νέας συμφωνίας. Η ανακοίνωσή μας επίσης τονίζει τη σημασία της ΙΚΑΟ και της IMO και αυτό νομίζω φαίνεται και από τις προτάσεις του εισηγητή. Δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά πόσο σημαντικές είναι οι δράσεις του IMO και της ΙΚΑΟ. Έχοντας εργαστεί πάνω στα θέματα αυτά και στο παρελθόν, μπορώ να σας εκφράσω και τη δική μας δυσαρέσκεια λόγω της καθυστέρησης ε, που έχουμε διαπιστώσει. Ωστόσο, αυτοί είναι οι διεθνείς οργανισμοί που ε, έχουν καθήκον να προωθήσουν την πολύπλευρη δράση. Πολύ σύντομα να αναφερθώ στο δικό μας όραμα όσον αφορά το Παρίσι. Η νέα συμφωνήση αποτελεί πολύ σημαντική ευκαιρία για μας για να έχουμε δράση που να ισχύει για όλους. Έτσι θα ξεφύγουμε από την παλιά ερμηνεία όσον αφορά τον καταμερισμό των ευθυνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει δηλαδή να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα όραμα για ε, μακροπρόθεσμο στόχο όσον αφορά την κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί στον τομέα των μεταφορών. Προβλέπεται μείωση μέχρι το 2005 σε σχέση με τα επίπεδα του 2010 που συνάδει απόλυτα με την ε, πέμπτη έκθεση αξιολόγηση ε, του ε, IPCC και αυτό είναι ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους που πιστεύουμε ότι ακολουθεί πολύ καλά την προσέγγιση μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Κοινοβούλιο για την ενεργό συμμετοχή του στην προετοιμασία της Συνόδου του Παρισιού. Σας ε, ευχαριστώ για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Βίρκουνεν. Yes, Mr. <laughs> Uh, Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρατηρήσεις σας. Περιμένω να λάβω την επόμενη εβδομάδα τις τροπολογίες σας και ελπίζω να έχουμε μια συνάντηση σύντομα μετά από αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών. Προσλέπω στη στενή συνεργασία με όλους σας. Ευχαριστώ πολύ. Μπας Eichhout. Ευχαριστώ πολύ και, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους και ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές. Θα συνεργαστούμε πάνω στις συμβαστικές τροπολογίες και οι τροπολογίες θα αποτελούν περισσότερο προσθήκη στη δουλειά που ήδη έχει γίνει. Μου άρεσε πολύ το θέμα που ανέφερε η Κριστίν. Θα χαρώ πολύ να προσθεθούν οι ε, τροπολογίες στην έκθεση και επίσης ε, το θέμα του Ήβο για την φορολογία και την αεροπλοεία. Είναι ενδιαφέρον το θέμα αυτό και θα δούμε πώς μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στην ε, γνωμοδότησή μας. Στον κόσμο Σλοτόφσκι να πω ότι συμφωνώ όσον αφορά τις υποδομές. Είναι σημαντικό αυτό. Όσον αφορά τις ε, διαφορές ανάμεσα στις χώρες, αυτό είναι σημαντικό θέμα και εντός του ΟΗΕ. Δεν μπορεί κανείς ε, να κάνει ούτε ένα βήμα χωρίς να ακούσει κανείς ότι πρέπει να είναι κοινή ευθύνη αλλά ε, διαφορετικά μοιρασμένη. Και θα ήθελα να τονίσω ότι και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις δικές μας πολιτικές υπάρχει διαφορά ε, ανάμεσα στο τι περιμένουμε ανάμεσα, από, από τα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δείτε και στη σχετική έκθεση ότι απαιτούνται ε, διαφορετικές ε, ε, προσπάθειες από τα διάφορα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει αυτό λοιπόν με τρόπο επαρκή και όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που οι στόχοι έχουν τεθεί λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και να αναφερθώ στην Ενεργειακή Ένωση, να δούμε τι μορφή θα έχει το κυβερνητικό τμήμα. Η Κομισιόν ε, εγκατέλειψε τις προσπάθειες εκεί, αλλά πτώση αυτό ήταν μια παρένθεση. Όσον αφορά αυτά που είπε ο Παβέλ, ναι, μια συνολική συμφωνία θα τα λάβει όλα υπόψη. Πολύ θα χαρώ να μην έχουμε ε, άλλη συζήτηση για το θέμα της ε, διαρροής ε, διοξιδίου του άνθρακα. Όσον αφορά την μονομερή δράση. Θα χαρώ πολύ να συζητήσω με την Γεζίνε, διότι εάν εξετάσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ήπειρο, εξαρτώμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Εάν μία χώρα θα πρέπει να περάσει πιο γρήγορα στη μετάβαση χωρίς να περιμένει τους άλλους, νομίζω ότι ε, η έγκαιρη δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και οικονομικά σοφή. Δεν θα θεωρούσα λοιπόν ότι είναι μονομερή σε δράση μόνο από κλιματικής πλευράς. Θεωρώ ότι είναι και μια οικονομικά σοφή κίνηση. Δεν ε, με εκπλήσει που κάποιος από τη Φιλανδία μιλάει για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι χρήσιμα αυτά και στον ε, ΠΙΤΑ και την ε, συζήτηση για τον καποτάζ. Θα πρέπει να είμαι ειλικρινής, δεν σκοπεύω να συμπεριλάβω αυτό το θέμα στην ε, έκθεσή μου, διότι θα συζητήσουμε πολλά θέματα στο Παρίσι, όχι όμως στο καμποτάζ. Νομίζω ότι ήδη έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε στο Παρίσι. Μία τελευταία παρατήρηση προς την Κομισιόν για τον IMO και την ICAO. Συμφωνώ ότι αυτοί οι διεθνεί οργανισμοί θα πρέπει να κάνουν τα επόμενα βήματα, αλλά... Νομίζω ότι το Παρίσι θα θέσει το πλαίσιο και τους στόχους για τους διάφορους τομείς. Βλέπω ότι αμφιβάλλετε λίγο. Θα πρέπει να μάθετε να κρατάτε πιο ουδετερή στάση να μην προδίδετε τα αισθήματα στην έκφρασή σα, αλλά αυτό, μπορούν να θέσουν τους δικούς τους ε, στόχους οι τομεί αυτοί και δεν έχουν πολλοί τομεί αυτό το προνόμιο. Να πω λοιπόν ότι εντός της Επιτροπής ΕΝΒΗ ζητήσαμε μία μελέτη, διότι αν κοιτάξουμε τους στόχους αυτούς ε, σε δύο φάσεις και τους τομείς της αεροπλοείας ε, και της ναυτιλίας, Ελπίζω το Παρίσι να σπρώξει τους οργανισμούς αυτούς, ε, ε, τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας ε, και την ΙΚΑΟ, να ξεφύγει από αυτήν την καθυστέρηση. Θα πρέπει στο Παρίσι να σπρώξουμε τους οργανισμούς αυτούς να πάρουν προς. Στην έκθεσή μου λοιπόν θα είμαι λίγο πιο φιλόδοξο στο θέμα αυτό από ό,τι άκουσα την Επιτροπή να είναι. Άκουσα, από όσα άκουσα από τους συναδέλφους έχω και την αίσθηση ότι θα υπάρχει πλειοψηφία υπέρ του να σπρώξουμε τους οργανισμούς αυτούς. Προσβλέπω στις επόμενες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ και για, την, για τις εκθέσεις και για ε, τις παρεμβάσεις σας. 5 ε, Ιουνίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και φτάνουμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε τους Ευρωπαίους συντονιστές ε, για τους ε, διάφορους ευρωπαϊκούς ε, διαδρόμους. Ε, ο Πέτερ Μπάλας δεν είναι παρόν, το ανέφερα ήδη αυτό. Έχουμε τον Κάρλο Σέκη, Ευρωπαίο Συντονιστή για τον διάδρομο του Ατλαντικού. Και ο Ματιό Γκρό μπορεί πολύ ευχαριστώ να έρθει στο βήμα, αν θέλει, αλλιώς μπορεί να παραμείνει στη θέση του. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Κάρλο.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 θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Μάρτιν Φούξ, νέο συνεργάτη στην Γραμματεία. Ε, μας προέρχεται από την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Νομίζω ότι θα συμβάλλει με την ε, πείρα του από εκεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή μας και προσλέπουμε στην καλή συνεργασία. Δίνω το λόγο στον Κάρλος Έκη. Thank you very much, ε, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, είμαι πολύ ευτυχής που είμαι σήμερα εδώ ε, για να συζητήσω μαζί σας. Να κάνουμε αυτή την αλλαγή ε, απόψεων για τον ε, διάδρομο του Ατλαντικού και προσβλέπω για τον οποίο είμαι συντονιστής και βεβαίως Έχω και ένα ωραίο ε, να σας δείξω. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να θεωρήσετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Ε, έχουμε στην περίοδο αυτή συνεργαστεί μαζί με τις διάφορες συνιστώσεις της διακυβέρνηση του διαδρόμου, ώστε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση του χρόνου και των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα σας κάνω μια σύντομη εισήγηση για το τι θα βρείτε στο έγγραφο και θα σας δείξω και κάποιες διαφάνειες. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ατλαντικού διαδρόμου. So the key features of Atlantic τα βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν του Ατλαντικού διαδρόμου είναι εδώ σε αυτό το πρώτο, στην πρώτη διαφάνεια. Καταρχήν έχει μια πολύ σημαντική συνιστόσα αναψυπλοεία, όπως βλέπετε και από την εικόνα και όπως λέει και το όνομα του διαδρόμου αυτού. Περιλαμβάνει 13 βασικά λιμάνια ε, τόσο θαλάσσια όσο και σε εσωτερικέ πλωτέ οδού και πολλά άλλα σημαντικά λιμάνια που ανήκουν στο συνολικό δίκτυο από την άποψη του ο σιδηροδρόμου, ο διάδρομος ε, ε, τέσσερα σιδηροδρομικών εμπορικών μεταφορών είναι η σπονδυλική στήλη και θέλω να τονίσω πως μόλις χθες η Γερμανία υπέγραψε την συμφωνία για να συμμετέχει στον ε, σιδηροδρομικό διάδρομο εμπορευματικών μεταφορών ε, αριθμών 4. Έχουμε λοιπόν τέσσερα διασυνοριακά τμήματα, δύο ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, ένα ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία και ένα ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Οπότε ε, συνδέει τρεις ε, πρωτεύουσες και έχει όμως κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, όπως υπάρχουν δύο ε, στην ε, δύο ε, στενά και μπορούμε να πούμε ότι ο Ατλαντικός διάδρομος συνδέει τον Ατλαντικό ωκεανό με πολύ σημαντικές χώρες δηλαδή και αγορές με την καρδιά της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό, την Κεντρική Ευρώπη. Ο ρόλος του θα είναι ακόμα πιο σημαντικός όταν θα διανοιχθεί η, ακόμη περισσότερο η διόρυγα του Παναμά και κατά συνέπεια θα επιτρέψει ακόμα μεγαλύτερη ροή προς την Ευρώπη μέσω του Ατλαντικού ωκεανού. Όπως μπορείτε να δείτε στο χάρτη, σε αυτή τη διαφάνεια που δεν είναι και πολύ ξεκάθαρη, αλλά εν πάση περιπτώσει φανταστείτε το λίγο, μαντέψτε λίγο. Ο διάδρομος είναι η κίτρινη γραμμή που πηγαίνει από την νότια Ισπανία και Πορτογαλία μέχρι το Μάνχαϊμ και το Στρασβούργο. Εδώ εστιάζουμε στις στα διασυνοριακά τμήματα, το σκούρο μπλε, είναι εκείνα τα διασυνοριακά τμήματα όπου γίνονται έργα κυρίως πάνω-πάνω ανάμεσα στην Γαλλία και τη Γερμανία εν μέρη στο, τη σύνδεση τη διασυνοριακή αφορά ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία και ε, επίσης για την Πορτογαλία συνεχίζονται έργα για την νότια σύνδεση στην Εύωρα, ενώ η βόρεια σύνδεση που υπάρχει από την Αβέιρα μέχρι τη Σαλαμάνκα λειτουργεί, αλλά χρειάζεται πολλές βελτιώσεις, για τις οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή μελέτες. Και θα αρχίσουν οι εργασίες στο εγγύς μέλλον. Στα δεξιά της διαφάνειας όλα τα αστέρια αντιπροσωπεύουν τις ε, αιτήσει που λάβαμε για καλά προγράμματα που έχουν υποβληθεί είτε στη διαγωνισμό που έγινε και έκλεισε το τελευταίο Φεβρουάριο, τον περασμένο Φεβρουάριο, είτε προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και βλέπετε ότι συμπεριλαμβάνονται τα περισσότερα σημαντικά λιμάνια, αλλά και άλλα σημαντικά projects που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση. Τώρα, αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα τέντη και τις τεχνικές ε, προδιαγραφές Σύντομα μπορώ να σας πω ότι λέει εκεί στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας ηλεκτροδότηση των σιδηροδρόμων, πολύ διευρυμένη, σχεδόν στο 90% αν και έχουμε τέσσερα διαφορετικά συστήματα ηλεκτροδότησης στην Ευρώπη. Πολλά πρέπει να γίνουν λοιπόν για να εισαχθούν κοινέ προδιαγραφές. Δύο διαφορετικές, ε, διαφορετικά ε, στενά όπου απαιτείται να έχουμε συμπεφωνημένο σχέδιο ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, ώστε να έχουμε σταδιακά επίλυση αυτού του προβλήματος. Για την ώρα η Ισπανία υψηλή ταχύτητα έχει προσαρμοστεί Όλα τα άλλα πρέπει να προσαρμοστούν. Η Επιτροπή σα εξάλλου πιστεύω ότι επισκέφθηκε την χώρα των Βάσκων τον περασμένο Μάρτιο και είδατε ποια είναι τα προβλήματα προς επίλυση συμπεριλαμβανομένων ε, των ε, πρόοδων που σημειώνονται στην περιοχή. Υπάρχει ισχυρή δέσμευση για επιτάχυνση της εισαγωγής όλων αυτών των σημείων και σημαντικό σημείο που συνδέεται με την προηγούμενη συζήτηση η ανάπτυξη της χρήσης του, φυσικού, του, του υγροποιημένου ε, αερίου στην αναψυπλοεία. συζητιέται εντόνως, είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και πρέπει να καλυφθούν και οι σχετικές ανάγκες λόγω της ACCA, δηλαδή τους, ε, τις ε, περιοχές ε, που συνδέουν την Βόρεια Αμερική με την Βόρεια Ευρώπη. Εδώ χρειάζεται να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί πόλοι, ε, φυσικά να γίνουν και επενδύσεις για τα πλοία. Οι μηχανές μπορούν να προσαρμοστούν για αυτό το στόχο και μπορούν να εφέρουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά το περιβάλλον, τη σημαντική συμβολή στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν είναι projects που είναι πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό τον διάδρομο. Και όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους, που βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση στον Ατλαντικό διάδρομο, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τα διαλειτουργικά συστήματα διοδίων για να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν αυτές τις ε, οδούς. Προτεραιότητες, λοιπόν, στόχοι μάλλον και προτεραιότητες, οι στόχοι είναι γνωστοί, η αύξηση της πολυτροπικότητας και η ισορροπημένη κατανομή στους διάφορους τρόπους μεταφοράς και ιδιαίτερα μεγαλύτερη χρήση των σιδηροδρόμων καθώς και του συστήματος των υποδομών, ιδιαίτερα για τις εμπορευματικές μεταφορές διαλειτουργικότητα, σύνδεση εθνικών δίκτυων, ανάπτυξη διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, χάρη στις λύσεις ε, ε, του προβλήματος των, ε, του ορισμού του ERTMS, του των διαφορετικών σιδηροδρομικών τροχιών και ούτω καθεξής. Και έπειτα ποιες είναι οι προτεραιότητες. Έχουμε την εξωτερική διάσταση προς τον Ατλαντικό, ωκεανό, την προώθηση της ναυσιπλοείας μέσω της καινοτομίας, της απλοποίησης, καθώς και των καθαρότερων ε, καυσίμων, όπως το υγροποιημένο αέριο η προτεραιότητά μας είναι να βελτιώσουμε την ε, σύνδεση μεταξύ των λιμανιών, την διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις υφιστάμενες πλατφόρμες, καθώς και τη σύνδεση με τους άλλους διαδρόμους που έρχονται σε επαφή με τον Ατλαντικό ε, διάδρομο, να εκπονήσουμε ένα κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης για να αλλάξουμε το σύστημα στο UIC ε, τον, το σύστημα των τροχιών, να συμπληρώσουμε τα τμήματα που λείπουν, έβορα Μέρδα και έβορα Παραντός, και να βελτιώσουμε τις αστικές ε, διελεύσεις, ε, να επιταχύνουμε τη χρήση του λιγροποιημένου αερίου καθώς και το εξυγχρονισμό των λιμένων. Έχει γίνει πολλή δουλειά στην Πορτογαλία, αλλά ακόμα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Και τέλος να αυξηθεί η ορατότητα του διαδρόμου, ώστε να μπούμε στις παγκόσμιες ροές, ε, για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις ευκαιρίες που προφέρονται. Αυτά είναι κατ' ουσίαν, ε, κύριε Πρόεδρε Κυρίες και κύριοι, τα όσα ε, περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή προτάσεις που μπορεί να έχετε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ζήτησαν το λόγο και ο Βίμ Φαντεκάμπ είναι ο τρίτος. Παρακαλώ. Ε, <clears throat> Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όσο περισσότερα μαθαίνω για τους διαδρόμους ε, του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, τόσο περισσότερο μου αρέσουν. Νομίζω ότι είναι τα πετράδια του στέματος της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών. Και η πολιτική μου ομάδα πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και να εντατικοποιηθεί. Χαίρομαι που βλέπω ότι το Στρασβούργο αποτελεί μέρος ενός διαδρόμου. Το TGV, το τρένο από το Στρασβούργο στο Παρίσι, μερικές φορές συναντά δυσκολίες ε, στο Σαβέρν. Ε, θα ήθελα να το πω αυτό στον ε, καθηγητή Ισέκη. Ελπίζω να μπορέσει να φροντίσει το τρένο να φτάνει στην ώρα του. Νομίζω ότι είσαστε υπερβολικά ευγενικό είστε σοφός άνθρωπος, αλλά εγώ θα ήθελα τα δομικά υλικά για να δώσω περισσότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, έχετε αρκετή χρηματοδότηση, θα τελειώσετε εγκαίρως, οι άδειε είναι εντάξει, η Ευρώπη δεν έχει χρόνο. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να επικρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να μου δώσετε τα εργαλεία για να κάνουμε τα πράγματα πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Είναι δύσκολο να μεταφερθεί η ενέργεια από το Μαρόκο στην Ισπανία και από την Ισπανία στη Γαλλία. Τα πυρηναία όρη μας εμποδίζουν. φαντάζεστε να υπάρξει κάποια σύνδεση εκεί. Αν μου πείτε ότι λέω ανοησίες, ε, μπορώ να το δεχτώ, αλλά έχετε εξετάσει τις δυνατότητες. Η Ενεργειακή Ένωση λειτουργεί. Ο κόσμος μπορεί να εκνευρίζεται με την Κομισιόν, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να συνεργαστούμε. Eh, Ευχαριστώ, κύριε Σέκη, για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Νομίζω ότι όλα αυτά που αναφέρατε είναι σωστά και συμφωνούμε με όλα αυτά. Συμφωνούμε, πιστεύω, η ευρεία πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Σε αυτά τα έργα σε αυτή την κολόνα τη στήλη που μας δείξατε στην ωραία σας διαφάνεια. Τα έργα που έχουν παρουσιάσει τα κράτη-μέλη για αυτόν τον άξονα τον Ατλαντικό που είχαν αστερίσκο. Είναι έργα που καλύπτουν τα δύο βασικά ερωτήματα που αναφέρατε εσείς. Δηλαδή οι διασυνοριακές περιοχές. Παρακαλώ συνάδελφε να κλείσετε το μικρόφωνο σας. Περιλαμβάνουν λοιπόν τα έργα αυτά τις διασυνοριακές ζώνες, γιατί εγώ για παράδειγμα ζω στη χώρα των Βάσκων και υποφέρομαι. Είμαστε διασυνοριακή περιοχή και υποφέρουμε από την κυκλοφοριακή συμφόρηση από χιλιάδες φορτηγά που περνούν από ε, τα εδάφη μας και δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει θέμα με το γαλλικό κράτος, το οποίο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το γεγονός ότι ε, η διασυνοριακή μετακίνηση είναι κάτι που πρέπει να έχει προτεραιότητα και πρέπει να την εφαρμόζει αυτή την προτεραιότητα αμέσως. Επομένως, ποια είναι η εικόνα σας για αυτά τα έργα με αστερίσκο, πώς θεωρείτε ότι διάκυνται οι τρεις χώρες που συνδέονται και τους αφορά αυτός ο Ατλαντικός άξονας, Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία. Και επίσης κλείνω λέγοντάς σας ότι πρόσφατα έχουν καταβληθεί κάποιες προσπάθειες. Η Ισπανική κυβέρνηση ως προς το κομμάτι που περνάει από τη χώρα των Βάσκων, το οποίο ονομάζεται το Βασκικό Ήψιλον, ε, μας λέει η Ισπανική κυβέρνηση ότι θα υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις ως προς την άφηξη των τρένων στις διάφορες πόλεις. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις επ' αυτού, γιατί ξέρετε σήμερα τον πρωί μιλήσαμε για τη Λευκή Βίβλο και για την ανάγκη συντονισμού και εκτέλεσης με αποτελεσματικό τρόπο και με προτεραιότητα εκτέλεσης των έργων, υλοποίησής τους. Και άρα ε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Οι προτάσεις, τα έργα που έχουν παρουσία στα κράτη-μέλη έχουν οριμάσει, είναι σε φάση Και να σας πω τέλος ότι μας λείπει, μας έλειψε ένα έργο, ένα σχέδιο που δεν παρουσιάστηκε για να έχει σχέδιο που αποσκοπεί να έχει περισσότερη συνοχή όλη αυτή η εφαρμογή του Ατλαντικού άξονα. Ευχαριστώ κυρία Καρίμα Ντέλη από τη Γαλλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε επιφορτισμένε με το καθήκον του συντονισμού για τον Ατλαντικό διάδρομο. Καταρχάς να σας ευχηθώ καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο διότι είναι προτεραιότητα ο αυτοκινητόδρομος και η σιδηροδρομική σύνδεση που προτείνεται, κυρίως για λόγους περιβαλλοντικούς, Δυστυχώς κρατώ την ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης με ημερομηνία 30 Απριλίου του 2015 όπου αναφέρεται ρητός ότι παρετούμεθα από την ύπαρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης από το Πάντο Καλέ μέχρι και το Λόντ που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2017 και που θα μετέφερε αυτό το τρένο 425.000 φορτηγά ε, το χρόνο. Ε, Αποσύριεται λοιπόν η γαλλική κυβέρνηση από την κατασκευή αυτής της σιδηροδρομικής μεταφοράς των φορτηγών. Ενώ είναι πολύ υποφελές το έργο αυτό και βεβαίως άπτεται της αρμοδιότητας του Ατλαντικού διαδρόμου πώς θα παραμείνουμε συνδεδεμένοι ενώ ο βασικός κορμός του έργου δεν θα υπάρχει γιατί δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη της Γαλλίας καταρχάς. Κατά δεύτερο, κάνατε διαπραγματεύσεις με τη γαλλική κυβέρνηση. Η γαλλική κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να το φτιάξει το έργο από τη στιγμή που πρέπει να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Και τρίτη ερώτηση ως προς την προόδο του, των εμπορικών μεταφορών, ε, των εμπορευμάτων μάλλον, ε, φρέτ, ε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε αυτό το διάδρομο τον Ατλαντικό. Ο κύριος Πάσκο. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Είχα καταλάβει ότι πιο αργά θα παρανέβαινε, θα παρενέβαινε ο κύριος Κάρλο Σέκη. Ωστόσο, θέλω να πω κύριε Πρόεδρε ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερο αυτός ο διάδρομος ο Ατλαντικός γιατί ε, εμπλέκεται εκεί η Ισπανία. Εκτιμώ ιδιαίτερο τον συντονιστή, είναι πολύ μελετημένος, είναι πολύ καλά καταρτισμένος, δεν θα πω διάφορα λόγια γενικόλογα, θα πάω στο ψαχνό. Θα σας ρωτήσω ποιες λύσεις προβλέπετε για προβλήματα τα οποία είναι αρκετά παλαιά ήδη. Κύριε Σέκη, λοιπόν, έρχομαι, στρέφομαι σε εσά και λέω, ξέρετε πολύ καλά ότι η Γαλλία δίνει προτεραιότητα στη σύνδεση μεταξύ Μπορντό και Λούζ, Μπορντό ε, και Τουλούζης. Ενώ τελικά ένας διάδρομος πρέπει να περνάει από διάφορες χώρες και το Μπορντό είναι κοντά στα γαλλοϊσπανικά σύνορα και η Τουλούζη. Λοιπόν, ποια προβλήματα εντοπίσατε ο συντονιστής και τι κάνετε για αυτά. Επίσης, το εύρος, το πλάτος της γραμμής στα τρένα υψηλής ταχύτητας στα ισπανικά έχει λυθεί το θέμα αυτό. Υπάρχουν δύο κριτήρια, η θέση της Κομισιόν και η θέση ισπανική που ε, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη ευελιξία στις περιφερειακές συνδέσεις. Θα φτάσουμε σε μια ε, μόνη λύση για διαλειτουργικότητα σε σχέση με το πλάτος της γραμμής ή μπορούν να συμβαδίσουν ε, διάφορα χαρακτηριστικά δικτύου, ε, διαφορετικά δίκτυα να, το πω έτσι. μιλάω για το κομμάτι το ισπανικό. Και δεν έχει λυθεί το θέμα της σύνδεσης Ισπανίας-Πορτογαλίας ακόμα. Πώς μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένες λύσεις, με ποιες προθεσμίες για τη μέριδα και τη σύνδεσή της. Και λείπει και το, η σύνδεση Αβέιρο Πορτογαλίας και Σαλαμάνκα Ισπανίας. Πώς αξιολογείται τα διάφορα πρότυπα εξηλεκτρισμού στο διάδρομο Και επειδή μιλάτε και πολύ καλά ε, ισπανικά, να σας πω ότι πιάνουμε το τάβρο από τα κέρατα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Άμεσα τέτα τέτα απευθεία σας τα θέτουμε με όνοματα επώνυμο. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και περιμένουμε την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Ο Παύλο Τέλιτσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή. Ναι. Ως συνέχεια στα όσα είπε ο Βίμ Βαντρικάμπ. Θα πρέπει να πω ότι όσον αφορά τις ε, πολιτικές τάσεις, νομίζω πως ε, το TNT ήταν η σημαντικότερη συμβολή στην κοινή πολιτική μεταφορών τα τελευταία χρόνια. Και Είχα την ευκαιρία να το παρακολουθήσω. Είναι ένα εξαιρετικό μέσο και έχουμε μια εξαιρετική ομάδα συντονιστών. Ε, ε, έχω να κάνω δύο ερωτήσεις που αφορούν τον ε, διάδρομο αυτών, τον άξονα αυτών, αλλά είναι γενικότερες φύσεις, όχι πολύ ειδικέ, γιατί δεν γνωρίζω σε κάθε λεπτομέρεια τον διάδρομο και ξέρω πως βρίσκεται σε καλά χέρια. Τι θα λέγατε Όσον αφορά τι οικονομικέ, τις δυνατότητες που έχουμε, λαμβάνοντα υπόψη ότι μόλι σήμερα το πρωί ο τριμερή ε, για το ΕΦΣΙ ολοκληρώθηκε και θα γνωρίζετε πολύ καλά ποιε είναι οι συνέπειες για το ΣΕΦ. Εσείς θα λέγατε ότι έχετε ήδη κάποιο είδος ανάλυση των επιπτώσεων ε, για όλους τους διαδρόμους, ιδιαίτερα ίσως για το δικό σας. Υπάρχει κάποια ανησυχία που μπορεί να έχετε ή όλα πάνε καλά. Η επιρροή θα είναι ίσως σχετικά μικρή. Εάν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις μπορείτε να μας πείτε αυτό. Γιατί θα πρέπει να έχετε κάποια εκτίμηση για το τι μπορεί να γίνει με την πρώτη, ε, το πρώτο, για τον πρώτο διαγωνισμό και ποιες θα είναι οι ανάγκες τα επόμενα χρόνια. Και σας ρωτώ για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει εμείς να λάβουμε κάποια θέση επί του αποτελέσματος και θα θέλαμε να λάβουμε τη σωστή απόφαση. Έχουμε λοιπόν φρέσκα στοιχεία. Θέλουμε να τα ξαναδούμε και πάλι, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε μια απόφαση Ε, σε σχέση με κάτι που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις ακριβώς επειδή κάποιοι θεσμοί δεν είχαν τη δημιουργικότητα και το θάρρος που χρειαζόταν. Ε, ξέρω ποια είναι η θέση της Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι ανεξάρτητη, πρέπει να, ε, φέρει αποτελέσματα και θα πρέπει να ξέρουμε γιατί δεν θα φέρει αν δεν φέρει. Ποιες είναι λοιπόν οι επιπτώσεις, πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε ή αν μπορούμε κάπως να σας βοηθήσουμε ως Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε στην επίσκεψή μας στην χώρα των Βάσκων, όπου διαπιστώσαμε ότι ναι, πράγματι θα υπάρχουν δύο διαφορετικά φάρδι των συνδρόμων. Δεν είναι δυνατόν να το αποφύγουμε αυτό. Το θετικό όμως στη χώρα των Βάσκων είναι ότι ελήφθη υπόψη ότι θα πρέπει να είναι κατάλληλες σειράγες για την μεταφορά εμπορευμάτων στην Γερμανία. Δεν το προσέξαμε αυτό και έτσι, οι Ισπανοί ήταν πιο έξυπνοι από ότι οι Γερμανοί. Το θέμα τώρα είναι πώς μπορούμε να ενώσουμε την Ευρώπη. Γαλλία λέει από το Πορδό μέχρι το σύνορο της Ισπανίας ε, δεν μας ενδιαφέρει πια. Ποια προγράμματα θα καταργηθούν. Η σύνδεση Λιών του δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 40 χρόνια και έχει στήχησει πάρα πολλά χρήματα ε, και με ένα κλάσμα αυτού του ποσού θα μπορούσαμε να ε, έχουμε την γραμμή από τον Πορντό στα σύνορα της Ευρώπης και θα ήταν μια χαρά ενωμένη Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν με την Κομισιόν, με τα κράτη-μέλη να συζητήσουμε τι είναι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δεύτερη παρατήρησή μου. Είπες ε, ότι η ενέργεια... Από... Α, νόμιζα ότι εσύ μου μίλησες όχι από εσά πήρα την ιδέα αυτή ότι είναι ανοησία. Α, όχι. Α, πρόεδρος, εσύ το επανέλαβες και εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν ανοησία αυτό. Φυσικά είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Χαίρομαι που ξεκαθαρίσαμε την ε, παρεξήγηση. Αλλά στην Ισπανία, στην ε, Νότια Γαλλία μπορούμε να ε, έχουμε ε, παραγωγή ηλεκτρικής ε, ηλιακής ενέργειας. Ε, δεν χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την ενέργεια από την Αφρική. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε τον μακρύτερο δυνατό αγωγό. Το θέμα είναι να έχουμε προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και για τον τομέα των μεταφορών. Σας δίνω το λόγο κύριε Σέκη για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας και τις παρεμβάσεις σας. Ε, ακούστηκαν διάφορες παρατηρήσεις, σας ξεκινήσω από το τέλος. Καταρχάς όμως να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά. Ποιος είναι ο στόχος αυτό του εγγράφου στο νέο κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Προβλέφθηκε το χρονοδιάγραμμα, έγινε διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, τις κυβερνήσεις κλπ. Ιδιαίτερα όμως αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μελέτης που έγινε και του λεγόμενου διαδρόμου 4 όπου είχαμε πάλι συνάντηση με όλους τους ενδιαφερομένους. Κάτι που συνέβαλε σε καλύτερη κατανόηση του θέματος ε, και καλύτερο εντοπισμό των αναγκών ε, προβλημάτων κλπ. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί. Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα. Δεν θα έχουμε όμως ποτέ ένα οριστικό πρόγραμμα εργασίας, διότι η διαδικασία αυτή είναι συνεχιζόμενη. Θα επικαιροποιηθεί του χρόνου και μετά σε δύο χρόνια πάλι. Αλλά οι διαβουλεύσεις θα ξεκινήσουν πάλι κατά τις ημέρες Διευρωπαϊκού Δικτύου στη Ρήγα, όπου θα καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα για τις μελλοντικές μας εργασίες. είναι κάτι το οποίο απαιτεί τη συμβολή όλων των ενδιαφερομένων για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη μου, στο έγγραφο αυτό απομένει ακόμα δουλειά να γίνει για να έχουμε έναν πολυτροπικό διάδρομο που να συνδέει με αποτελεσματικό τρόπο τις τέσσερις χώρες και που να συμβάλλει σε μια πιο ενοποιημένη εσωτερική αγορά. Δεν είναι λοιπόν απλά απεριθμισή ονείρων. Απαιτούνται βέβαια πολλοί πόροι για να γίνει αυτό. Πρόοδος πραγματοποιείται, αλλά πιο αργά από όσο ελπίζαμε, λόγω έλλειψης ε, πόρων, λόγω της κρίσης κλπ. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, το βασικό πρόβλημα είναι οι πόροι. Όπως σίγουρα όλοι γνωρίζετε, λάβαμε σημαντικό αριθμό πολύ καλογραμμένων προγραμμάτων ναι, τα οποία περιέγραφαν τι απαιτείται. Δεύτερον, αποτελεί απάντηση σε όσους λένε ότι δεν υπάρχουν αρκετά προγράμματα. Θα είναι δυνατόν να καλύψουμε μόνο το 1 τρίτο της ε, συγχρηματοδότησης. Ο συνολικός όγκος των επενδύσεων λοιπόν ξεπερνάει κατά πολύ τα 12 δισεκατομμύρια. Πετύχαμε λοιπόν μία συμφωνία, αυτό είναι θετικό, όλοι είναι ικανοποιημένοι με τον συμβιβασμό. Τώρα θα θέλουμε να τον εξετάσουμε αναλυτικά, να μας πείτε κι εσείς αν σας ικανοποιεί. Τουλάχιστον απελευθερώνονται κάποιοι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν στο εγγύς μέλλον ε, σε επόμενο γύρο υποβολή προσφορών. Ανοίγουν όμως όλα αυτά το δρόμο για το λεγόμενο σχέδιο Juncker. Η κυρία Μπιλπάο αναφέρθηκε στα ε, καλύτερα προγράμματα τα οποία ε, μπορούν ε, να ταιριάξουν καλά με την προσέγγιση Juncker. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα λυθούν τα προβλήματα αυτά. Η Γενική Διεύθυνση MOVE ε, ασχολείται με το θέμα αυτό. Εγώ, ο κύριος Πότεφικ και ο κύριος Κρίστοφ συμμετείχαμε σε διάλογο πάνω στο θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε. Το βασικό λοιπόν είναι οι πόροι. Πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους ε, προς όφελος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα προγράμματα αυτά για να εξαλείψουμε τα εμπόδια. Όταν ολοκληρωθεί η δουλειά αυτή θα είμαι πολύ ικανοποιημένος και θα χαρώ πολύ να έχω περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Να απαντήσω σύντομα σε αυτά που μας είπατε. Ε, τα σημείωσα και θα τα εξετάσουμε αναλυτικά. Αυτό που συμβαίνει όμως τώρα είναι ότι οι κυβερνήσεις ε, και όχι μόνο αυτές ε, στον διάδρομο αργούν ε, να τηρήσουν ε, τις υποχρεώσεις τους. Τηρούν βέβαια τη συμφωνία, το οποίο είναι θετικό. Γίνονται μελέτες και θα επιταχύνουν οι εργασίες στο εγγύς μέλλον για να καταλήξουμε σε ικανοποιητική συμφωνία με την Ισπανία προς όφελος ε, και της Ισπανίας, η οποία έχει επενδύσει πολλά στο θέμα αυτό. Είμαι αισιόδοξο λοιπόν ότι αυτό το μέρος του διαδρόμου, όπως και το Ίγκαβέρο Σαλαμάνκα, που είναι σημαντικό πρόγραμμα, θα υποβληθεί σύντομα από την Πορτογαλία και ότι έτσι θα έχουμε καλή ανάπτυξη. Λυπήθηκα λίγο με την ε, αναβολή του αυτοκινητόδρομου Ελπίζω ότι η απόφαση αυτή θα επανεξεταστεί στο εγγύς μέλλον. Είμαι πολύ ευαίσθητος απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα, την ε, συμφόρηση στη χώρα των Βάσκων αλλά και σε άλλα μέρη. Ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από τα προβλήματα αυτά, διότι αλλιώς θα καταλήξουμε σε τεράστια αντίφαση. Θέλουμε περισσότερες ε, ναυτοπλοϊκές ροές στον ε, Ατλαντικό διάδρομο, από την άλλη όμως θέλουμε να αποφύγουμε τη συμφόρηση. Η μόνη λύση λοιπόν είναι να βελτιωθεί η μεταφορά εμπορευμάτων με σιδηρόδρομο. όταν θα είναι διαθέσιμη αυτή η υποδομή και όταν δοθούν τα σωστά κίνητρα στους οικονομικούς φορείς και όχι όπως τώρα που δίδονται ε, σε λάθους φορείς ε, τα κίνητρα, θα λυθούν τα προβλήματα αυτά. και δεν θα έχουμε μείωση των εμπορικών ροών. Θα μπορέσουμε να τις αυξήσουμε σεβόμενοι και το περιβάλλον. Απαιτούνται όμως επενδύσεις και βούληση. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, να σας πω ότι μιλώ πολύ ανοιχτά, πολύ ειλικρινά Σημαντικό είναι να υπάρχει η βούληση, υπάρχει ευρεία συνένεση ότι αυτά πρέπει να γίνουν. Ε, υπάρχουν επιφυλάξεις λόγω οικονομικών προβλημάτων, διότι αν δαπανίσει κανείς ένα εκατομμύριο εδώ, λείπει από κάπου αλλού. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Και όπως έχουν δείξει πολλές μελέτες στο θέμα αυτό. Τα χρήματα που δαπανώνται για σωστές υποδομές όχι μόνο έχουν δαπανηθεί με σωστό τρόπο, αλλά συμβάλλουν θετικά στο ΑΕΠ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θέλετε περισσότερες πληροφορίες και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας στην κοινή μας προσπάθεια.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 ich Καλωσορίζω τώρα θερμά τον Ματιέ Γκρός που είναι γνωστός σε όλους μας ε, γιατί μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν Ευρωβουλευτής μέλος της Επιτροπής μας. Τώρα είναι συντονιστής για τον διάδρομο Μέσης Ανατολής ε, Ανατολικής Μεσογείου. Δέκα λεπτά έχει χρόνο ομιλίας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως σας είπα, σήμερα θέλω κυρίως να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Σύντομα όμως για τον ίδιο τον διάδρομο. Εννέα κράτη-μέλη αφορά ο διάδρομος αυτός. 15 κόμβους έχουμε, 15 αεροδρόμια λιμάνια, 12 λιμένες και θέλαμε να συγκρίνουμε αυτά που έχουμε στις κατευθυντήρες γραμμές και αυτά που ισχύουν για το διάδρομο. Στην επόμενη διαφάνεια λοιπόν βλέπετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο διάδρομο αυτό. η ηλεκτροδότηση, το βάρος ανά άξονα, το μήκος των τρένων. Βλέπετε εδώ ποιες θα είναι οι προκλήσεις τα επόμενα χρόνια για αυτόν τον διάδρομο και ποια θέματα θα πρέπει να τονίσουμε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές. Ε, αν πάρω το τρένο στο Αμβούργο και θέλω να πάω στην Αθήνα, τι γίνεται, αυτό εξετάσαμε. Εφτά διαφορετικά ε, συστήματα ασφαλείας έχουμε. Συνολικά τρεις διαφορετικές τάσεις. Τέσσερις φορές πρέπει να αλλάξουμε ε, τη μηχανή του τρένου. Μέγιστο μήκος 600 μέτρα, γνωρίζοντας ότι στη Βουλγαρία σε κάποια μέρη ε, Έχουμε μικρότερο μήκος, ε, έχουμε μέγιστο βάρος, ε, μέγιστη ταχύτητα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στους σιδηροδρόμους να ποντάρουμε στην διαλειτουργικότητα. Και για να σας δώσω πιο συγκεκριμένη η εικόνα. Σας δείχνω εδώ διάφορους χάρτες. Βλέπετε καταρχάς το βάρος ανά άξονα. Ε, στην πράσινη γραμμή τα πάμε καλά, στην κόκκινη όχι. Αυτό δείχνει την ε, έλλειψη συνοχής στο σύνολο του ε, διαδρόμου. Μίλησα για το μήκος των τρένων στην Γερμανία. Αρκεί, αλλά όσο πιο νότια πάμε και με διαφορά ανάμεσα στην Πρατισλάβα και νότια της Βουδαπέστης, αυξάνεται το πρόβλημα του μήκου των τρένων. Στην Ελλάδα λύνεται εν μέρη το πρόβλημα αυτό. Κατόπιν έχουμε την εσωτερική ναυσιπλοεία. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Βλέπετε όμως και εδώ τις προκλήσεις στην διαφάνεια. Βλέπετε το βάθος που απαιτείται για να έχουμε πλωτότητα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι πολύ σημαντική η πρόκληση αυτή. Γενικά, λοιπόν, στον διάδρομο αυτόν είναι σημαντικό να τονίσουμε τη διασυνοριακή διάσταση. Είναι πολύ σημαντικά εδώ κάποια διασυνοριακά προγράμματα και δουλειά μας ε, είναι να φέρουμε τους ανθρώπους ε, κοντά ε, από τις διάφορες χώρες για να συνομιλήσουν ανάμεσα στην Πράγα, την Αυστρία, την Ουγγαρία ανάμεσα στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα επίσης. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα θέματα. Δεύτερον, στον βορρά του διαδρόμου, στο Αμβούργο και στην Βρέμη, έχουμε μεγάλα λιμάνια, τα οποία λειτουργούν όμως μόνο αν λειτουργεί και η γύρω περιοχή. Στο Αμβούργο έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και για τα κοντέινερ τον μεγαλύτερο. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολυτροπικό σύστημα για να ε, ανακουφίσουμε από κάποια βάρη τον λιμένα αυτόν. Αυτό λοιπόν σχετίζεται με τη συνέχεια του διαδρόμου. Στο σύνολο του διαδρόμου μας ενδιαφέρει η πολυτροπικότητα, η ε, σχέση ανάμεσα στα διάφορα ε, είδη μεταφορών. Αναφέρθηκαν οι επενδύσεις. Ε, αξιολογήσαμε περίπου τον όγκο των μεταφορών, 47 δισεκατομμύρια. Υπολογίζουμε λοιπόν περίπου 50 δισεκατομμύρια, αλλά τα 25 δεν ε, προβλέπονται ακόμα στη χρηματοδότηση. Αυτό είναι μια πολύ χοντρή αξιολόγηση. Γνωρίζετε τα νούμερα, ξέρετε τι έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι αυτά που έχουμε αποφασίσει στις κατευθυντήριες γραμμές του διευρωπαϊκού δικτύου θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας για να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια. Αυτά που κάνουμε εμείς οι συντονιστές μαζί με τις 27-28 διορθώνει ομιλητής ε, χώρες σε άμεσο διάλογο αυτά οδήγησαν στο να έχουμε πάρα πολλά προγράμματα, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε όριμα προγράμματα. Εμείς μπορούμε μόνο σε έναν ε, διάδρομο να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους ε, της διευκόλυνσης ε, συνδέοντας την Ευρώπη. Πιστεύω ότι με πολλά μικρά προγράμματα μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε αυτόν τον διάδρομο και αυτό θα ήθελα να το τονίσω. Εδώ βλέπετε απάντηση στο θέμα πώς έχουν τα οικονομικά. Περιμένουμε μια δεύτερη διευκόλυνση ε, συνδέοντας την Ευρώπη. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του διαδρόμου αυτού. Τις έχω απαριθμίσει εδώ, δεν θα σας τις αναγνώσω αλλά θα ήθελα να τονίσω ένα ή δύο πράγματα. Εντός ε, του διαδρόμου ε, έχουμε τονίσει τη διασυνοριακή λειτουργία. Δεύτερον, ε, την εσωτερική ναυσιπλοεία, η οποία όμως γενικά αποτελεί δύσκολο πρόβλημα και επίσης την ανακούφιση των λιμένων με χρήση των σιδηροδρόμων. Επισκεφτήκαμε τη Δρέσδη, την Πράγα, ε, το Αμβούργο, την Βρέμη. Διαπιστώσαμε ότι η αδυναμία της εσωτερικής ναυσιπλοείας ε, οδηγεί ήδη τώρα σε υπερβολική επιβάρυνση των σιδηροδρόμων. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Γερμανία και η Τσεχία να ασχοληθούν από κοινού με ε, τον Έλβα και να δοθεί σαφής απάντηση και σημαντικό για μένα είναι ο ποταμός ε, Έλμπε είναι προτεραιότητα για μας ή όχι. Ε, αν ναι θα πρέπει να λάβουμε σαφή απόφαση και αν η απάντηση είναι όχι τότε δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε περαιτέρω. Είναι πολύ ε, απλή αυτή η ερώτηση, είναι πολύ σαφής η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί. Επίση πραγματοποιούνται εδώ μεταφορές οι οποίες δεν μπορούμε να πραγματοποιηθούν στο δρόμο ή στους σιδηροδρόμους. Νότια του Αμβούργου προς ε, την Δρέσδη υπάρχουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Εάν δεν υπάρξουν ε, εξελίξεις αυτό θα είναι προβληματικό για αυτές τις επιχειρήσεις. Και περιμένουμε μία ε, μελέτη σχετικά με τις θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν. Με το διευρωπαϊκό δίκτυο θέλουμε να έχουμε ένα ενιαίο σύνολο. Όσον αφορά τον ποταμό Έλβα, ιδιαίτερα στην Πράγα και στην Δρέσδη υποβάλαμε πρόταση να υπάρξουν ε, επαφές όχι μόνο στον τομέα ε, των μεταφορών και των πολιτικών, ε, αλλά και σε επίπεδο μη κυβερνητικών οργανώσεων, ώστε να αναλυθεί η κινητικότητα σε αυτές τις περιοχές διότι δεν θέλουμε απλά να παρουσιάσουμε ως δύσκολο έναν τρόπο μεταφορών, εάν, χωρίς να έχουμε εξετάσει τις εναλλακτικές λύσεις στους σιδηροδρόμους και τις οδικές μεταφορές. Αν οδηγήσει κανείς από τη Δρέσδη μέχρι την ε, Πράγα θα διαπιστώσει ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, οι σιδηρόδρομοι είναι, ε, τα τρένα είναι πλήρη είναι γεμάτα και θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτή λοιπόν είναι η μέθοδος που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Στην Ρήγα υποθέτω θα έχουμε μία συνάντηση Και αυτό σημαίνει ότι πάλι αναδιάδρομο θα συναντηθούμε με τους εταίρους, όχι μόνο με τους υπουργούς, αλλά και τους περιφερειακούς εταίρους και τους εκπροσώπους των σιδηροδρόμων κλπ. Τελευταία παρατήρηση όσον αφορά την χρηματοδότηση. Ε, ξέρω ότι τη νύχτα έγινε τριμερής ε, διάλογος, ε, αλλά ο διάδρομος πάνω στον οποίο εργάζομαι εγώ έχει το πλεονέκτημα ότι εκτός από τη Γερμανία έχει να κάνει αποκλειστικά με κράτη του Ταμείου Συνεχής, το οποίο σημαίνει ότι και φέτος και του χρόνου θα μπορέσουμε να ε, έχουμε μία πρόσκληση υποβολής προσφορών. Μέχρι το 2017 έχουν καθοριστεί τα ποσά αναχώρα. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά θα έχουμε λιγότερα προβλήματα όσον αφορά την κατανομή των πόρων, διότι οι χώρες γνωρίζουν πώς θα γίνει η κατανομή των 11 300 εκατομμυρίων. 7 δισεκατομμύρια διατίθενται για τον διάδρομο αυτό. Και είναι σαφή οι οδηγίες ότι μέχρι το 2017 μπορούν να απορροφηθούν αυτοί οι πόροι. Σύμφωνα με την αρχή, use it or lose it. Ε, πρέπει να απορροφηθούν, αλλιώς χάνονται οι πόροι αυτοί. Αυτά για τον διάδρομο αυτόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ, Ματιό Γκρός. Ο Βιμ Φαντεκάμπ. Πρόεδρε, εκ νέου και για τελευταία φορά σήμερα σας ευχαριστώ ειλικρινά να θυμίσω την ε, παρατήρησή μου για το κοσμήματο του θέματος. Όταν το βλέπει κανείς όλα αυτά, παίρνει ενέργεια, παίρνει, ενθουσιάζεται. Το τι είναι δυνατόν να γίνει στην Ευρώπη είναι υπέροχο. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για προβλήματα. Εδώ πραγματικά με γεμίζει ενέργεια και ενθουσιασμό όταν να μιλάμε για ένα τέτοιο διάξονα. Είναι διαφορετικά δε τα όσα μας λέει ο κύριος Κρός. Ξέρει καλά το παιχνίδι και πάει κατευθείαν στο στόχο. Ε, τα λέει πιο δυναμικά από τον καθηγητή Σέκη. Ε, όχι, τα λέω εγώ έξω από τα δόντια. Πρέπει να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Ε, είπατε ότι έχουμε αρκετά χρήματα. Και η αρχή είναι χρησιμοποίησέ τα, αλλιώς θα τα χάσεις. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πρόβλημα στην Ευρώπη όταν μιλάμε για άδειε. Το δεύτερο πρόβλημα που αφορά το FC, το FC αν όλα πάνε καλά θα δώσει χρήματα στα αεροδρόμια. Για τα λιμάνια και για τους σιδηρόδρομους θα είναι πιο δύσκολο. Η ΕΤΕΠ συνεργάζεται ή όλα γίνονται μέσω της Κομισιόν. Ποιες είναι οι σχέσεις. Μπορείτε να δημιουργήσετε τέτοιου είδους ε, συνεργασίες για να έχετε περισσότερα χρήματα. Και έπειτα, η προσοχή στην Κίνα. Να μένονται επενδύσεις από τους Κινέζους για τη σύνδεση ανάμεσα στη Βουδαπέστη και το Βουκουρέστι. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε αυτόν τον άξονα και την Κίνα. Και τέλος, ξέρω πως δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά αυτός ο άξονας είναι ένα, λείπει ένα μικρό κομματάκι για να φτάσει κανείς στην Κωνσταντινούπολη. Ε, μια μικρή προσπάθεια χρειάζεται. Τι πιστεύετε εσείς. Πήγαμε στη χώρα των Βάσκων ε, και μαζί με τον Ερτού και άλλους πήγαμε και στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί γίνονται πολλά πράγματα. Και τέλος, σε σχέση με τον καθηγητή ΣΕΚ, όλες αυτές οι επενδύσεις δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει να το πούμε ότι μπορεί να κουβεντιάζουμε όσο θέλουμε για βιωσιμότητα, για ε, ποδήλατα, αλλά πρέπει και να δουλέψουμε, να μην μιλάμε μόνο για ποδήλατα. Ευχαριστώ, θα το σχολιάσω αργότερα. Σαγιάλα Σέντερ. Σχεδόν απειλητικό ακούγεται αυτό. Τέλος πάντων, να ευχαριστήσουμε θερμά τον συνάδελφο κύριο Ματιό Γκρόσο για τον ενθουσιασμό. Για, την, ε, για το συντονισμό του σε αυτό τον πολύ περίπλοκο διάδρομο με τις τόσες δυσκολίες και αυτή είναι και η μεγάλο, μεγάλη πρόκληση. το σωστό είναι να έχουμε δια, διαδρόμους σε όλες τις επικράτειες, σε όλες τις περιοχές και όχι σε ορισμένες. Μακάρι και κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, βάσει του σχεδίου του Πρόεδρου Γιούνκερ, προβλέπει και δίνει δυνατότητες ρεαλιστικές Θα ρωτήσω και τον κύριο Κάρλο Σέκυρη Δημερός να μου τις εξηγήσει. Όμως, ε, ρωτώ εσάς κύριε Γκρός, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το νέο εργαλείο ε, εδώ για το θέμα μας. Να μην ε, μετατρέψουμε το συνδέοντας την Ευρώπη, το Connecting Europe, σε μέρος του ΕΦΣΥ. Να μην απλά δηλαδή με το ονοματίσουμε, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι ένα σημαντικό μέρος των πολύ μεγάλων έργων να υλοποιηθεί με αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο ή εργαλείο. Και πρέπει να δείξουμε σε όσους εμπλέκονται στον τομέα των μεταφορών ότι πράγματι το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, μπορεί να αξιοποιηθεί και για τις μεταφορές και θα αξιοποιηθεί και για τις μεταφορές. Σήμερα άκουσα ότι το ΕΦΣΙ θα ασχοληθεί με τη βιομηχανία, με την ενέργεια και ούτω καθεξής. Άρα, σας χρειαζόμαστε, εσάς που γνωρίζετε ε, το θέμα της απασχόλησης, των μεταφορών, του πώς όλα αυτά βοηθούν στην οικονομία, να μας βοηθήσετε για να προωθήσουμε τις μεταφορές, να εντοπίσουμε έργα σε κάθε διάδρομο που θα μπορούσε να ήταν επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και αυτό να το διεκδικήσουμε μέχρι θανάτου. Να είναι βέβαια καλύτερα, μπορεί να γίνουν ή χειρότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει να διεκδικήσουμε μέχρι τελική πτώσεως να υπάρχει χαρτοφυλάκιο μέσα στο ΕΦΣΥ έργων μεταφορών. Ευχαριστώ. Ο Παύλο Τελίτσκα. Ναι, ένα τελευταίο κομμάτι τσεχικής ε, διπλωματίας. Έχει φανεί ότι θα είστε στο μέλλον εξαιρετικό συντονιστής, ε, ε, συνάδελφε από τις κάτω χώρες. Ωστόσο, ο διάδρομος αυτός με αφορά πολύ περισσότερο και χαίρομαι ιδιαίτερο με την παρουσίαση αυτή. Θα μιλήσω για την πλευσιμότητα του ΕΛΜΠΑ. Θα μπορούσε κανείς πολύ δύσκολα να τα κάνει χειρότερα από ό,τι οι στο παρελθόν. Δεν είχαμε προτεραιότητες, δεν υπήρχε σαφής πολιτικός ε, ρόλος, ε, κατεύθυνση, δεν ήξερε η δεξιά τι είπε η αριστερά και αντιστρόφως. Έχουν αλλάξει αυτά με τον Υπουργό Μεταφορών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και πιστεύω ότι πέρα από την γερμανοτσεχική διάσταση στην οποία αναφερθήκατε είναι θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί, υπάρχει και μια άλλη διάσταση στο θέμα. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, οι συνάδελφοί σας ίσως γνωρίζουν περισσότερα. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για κάποιες περιβαλλοντικές πτυχές γύρω από το Μίλνικ και Χρειαζόμαστε να αναλάβουμε δράση λίαν συντόμως. Ίσως η DG MOVE και η DG ENVY ε, από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην έχουν τον απαραίτητο συντονισμό που χρειάζεται. Δεν μπορεί κανείς να είναι κάθε δεύτερη εβδομάδα στην Πράγα. Ωστόσο, να υπάρχει συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών Περιβάλλοντος ΣΥΝ ΜΚΟ. Ε, είναι πολύ σοβαρό το χρονοδιάγραμμα και είναι, καλός, ε, είναι καλές οι θετικές σκέψεις από πλευρά σας. Είναι καλό να προβληθούν, να φανεί η συνολική άποψη. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις με τους εκτελεστικούς διευθυντές και με τους εταίρους πρέπει να συναντηθούν οι δύο υπουργοί, κυρίως ο Υπουργό Μεταφορών, δεν έχουν αναλάβει καθήκοντα εδώ και πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβουν τις ΜΚΟ. Ο χρόνος κυλάει και θα πρέπει να ληφθεί μια κάποια απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω βάλει και το δικό μου όνομα στον κατάλογο των ομιλητών. ανέφερε στην προτεραιότητα των διασυνοριακών προγραμμάτων, αλλά και τα μικρά προγράμματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια μεγάλη στροφή όσον αφορά την προσέγγιση μας και τις πράξεις μας. Δεύτερον, είπε ότι είναι πολύ σημαντική η υποδομή γύρω από τους λιμένες στο Αμβούργο πολλά εμπορεύματα, τα περισσότερα από τα πλοία περνούν ε, στους σιδηροδρόμους μετά. Αυτό μας δείχνει ότι γίνεται. Και τρίτον έχουμε το θέμα της εσωτερικής ναυσιπλοείας και του ΕΛΒΑ που αναφέρθηκε. Ποια λοιπόν είναι τα γεγονότα. Τα τελευταία 20 χρόνια η εσωτερική ναυσιπλοεία στην Ευρώπη ε, έχει μειωθεί από το 20% στο 8%. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει υποδομή, οφείλεται στο ότι η εσωτερική ναυσιπλοεία είναι πολύ αργή και είναι πολύ αραιό το δίκτυο και γι' αυτό έχουν πλεονεκτήματα οι άλλοι τρόποι μεταφορών. Τι διαφορά κάνει αυτό, μπορώ να σας το πω. Ε, πριν 30 χρόνια από το Ίγκοστατ στην Μαύρη Θάλασσα έπρεψα στον Δούναβη και ε, σχεδόν κάθε 10 χρόνια ε, έπρεπε, με, το κουπί πήγαμε και έπρεπε κάθε 10 λεπτά να κάνουμε στροφή λόγω των κυμάτων. Ε, πρόσφατα έκανα πάλι την ίδια διαδρομή, τρία σκάφη είδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλο ο Δούναβη, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλοία. Όλες οι χώρες όμως ονειρεύονται αύξηση της ναυσιπλοείας όταν έχουμε την υποδομή, αλλά δεν θα την έχουμε. Στο Βερολίνο είδαμε ότι έγιναν έργα για την εσωτερική ναυσιπλοεία στο στον ε, λιμένα. Τα χρήματα βέβαια ήρθαν από την ε, Ομοσπονδία της Γερμανίας, ευχαριστώ στα πήραν τα χρήματα, αλλά τίποτα δεν άλλαξε αυτό. Ε, μετά έχουμε το κανάλι Ειρηνού Δούναβη. Αυτό επρόκειτο να είναι μεγάλη επένδυση. Και το 1980 με 82 θεωρήθηκε ε, η μεγαλύτερη ανοησία αυτό το κανάλι μετά τον πύργο της Βαβέλ. Το μόνο θετικό είναι ότι είναι πολύ ωραία διαδρομή, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει και με πολύ πιο οικονομικά μέσα. Ο ωραίος ποδηλατόδρομος που υπάρχει εκεί. Στη Γερμανία λοιπόν υπάρχει μεγάλο δυναμικό λόγο της προστασίας ε, το, του περιβάλλοντος. χτίστηκε νέος λιμένας ε, στον ε, Έλβα. Ε, έγιναν έργα στον Έλβα μόνο μέχρι το Αμβούργο. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσεις. Κατά μήκο του Έλβα υπάρχει πολύ ωραία σύνδεση σιδηροδρομική, η οποία όμως δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένη. 25 χρόνια χρειαζόμασταν για να καταστρώσουμε το σχέδιο, το οποίο ακόμα δεν εφαρμόστηκε. Λέμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, αλλά τα εμπορεύματα σε αυτόν τον διάδρομο θα μπορούσαν κάλλιστα να ε, μεταφερθούν με το σιδηρόδρομο, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα ε, έργα και γύρω από την Δρέσδη. Θα πρέπει λοιπόν να λάβει κανείς πρώτα την απόφαση να δώσουμε πλεονεκτήματα στον σιδηρόδρομο, να γίνεται έτσι η μεταφορά των εμπορευμάτων, να είναι αυτή η προτεραιότητά μας. Και εάν δεν αρκεί αυτό, μπορεί κανείς να σκεφτεί περαιτέρω τι θέλει να κάνει, αλλά τυφλά μετά από 20 χρόνια Και με τέτοια απώλεια της εσωτερικής ε, ναυσιπλοείας στην Ευρώπη δεν μπορεί κανείς να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Ε, εάν ε, κατεδαφίσει κανείς το Eurocenter στις Βρυξέλλες και το ανοικοδομήσει, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Έχει όμως νόημα κάτι τέτοιο νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες ιδέες που υπάρχουν. Γιατί είναι τόσο σημαντική η εσωτερική ναυσιπλοεία. Στη Γερμανία έχει γίνει στην μελέτη ε, δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας στην διοίκηση. Προσοχή λοιπόν όταν ε, μιλάμε για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Φυσικά θέλω να καταπολεμήσουμε την ανεργία, ε, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό με λογικά έργα. Ματιό Εγκρός, έχεις πάλι τον λόγο για να απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υποθέτω ότι δεν ήταν ερώτηση, ήταν ε, δήλωση αυτά που μας είπατε. Ε, ναι, φυσικά έχω μια ερώτηση, λέει ο πρόεδρο. Ποια είναι η γνώμη σα. Ε, ο κύριο Γκρό, ναι, θα μπορούσα να σα εξηγήσω ποια είναι η γνώμη μου. Πάντω, όταν βλέπω συνολικά τον διάδρομο αυτόν, και όταν μέχρι τέλη Ιουνίου θα δούμε τις οικονομικές συνέπειες και τις Θέσει απασχόληση που θα δημιουργηθούν. Δεν θα μιλάμε πια για επένδυση δισεκατομμυρίων, θα μιλάμε για ε, δημιουργία δυνατοτήτων και δεν θέλουμε να αποκλείσουμε ε, τρόπους μεταφορών. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τη σχέση ανάμεσα στην οικονομία και την οικολογία. Δεν νομίζω όμως ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συνδυαστεί. Στην Πράγα ε, συναντήθηκα με τους υπουργούς και στην Δρέσδη και μου είπαν ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και να δούμε τι πρέπει να γίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα στον Έλβα. Ε, θα πρέπει ε, να έχει 365 ε, μέρες το χρόνο βάθος 1,60, αλλά μόνο 40 μέρες το χρόνο έχει τέτοιο βάθος. Για το 1 τρίτο του χρόνου, λοιπόν, ο ο ε, οικονομικός φορέας δεν ξέρει αν μπορεί να μεταφέρει από εκεί τα εμπορεύματα. Αυτό λοιπόν είναι φαύλος κύκλος. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε ποιες είναι οι ελλακτικές λύσεις. Όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, ε, συμφωνώ κατά 100%. Αλλά πήγαμε και στη Βρέμη, που είναι απίστευτο σημείο συμφόρησης ε, για τους σιδηροδρόμους. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλοία που φτάνουν στους λιμένες με χωρητικότητα 80 με 100.000 ε, ε, τόνους, ε, αλλά θα πρέπει και η γύρω υποδομή να αντέχει αυτούς τους όγκους. Από την Σεχία και από άλλες χώρες του διαδρόμου έχουμε εμπορεύματα για τον Βορρά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να είναι διασυνοριακές οι λύσεις. Ε, νομίζω ότι τα προβλήματα δεν είναι καθαρά γερμανικά, είναι ε, προβλήματα που αφορούν τη σύνορα του δρόμου και τουλάχιστον έξι χώρες θα πρέπει να έχουν λέγη. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το περιβάλλον, αλλά θέλω να πάρω το πλοίο. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να είναι ανοιχτέ προς συζήτηση και γι' αυτό είχα και τη συνάντηση με τους υπουργού. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει απλά να αρχιοθετήσουμε το θέμα του διαδρόμου και της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δεύτερον, συνεργασία ανάμεσα στην Γερμανία και στη συγκεκριμένη περίπτωση την Τσεχία. Θέλαμε μια μορφή διασυνοριακής συνεργασίας, να εξετάσουμε δομές που υπάρχουν σε άλλα μέρη και τα μέρη να συναντηθούν και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Θα πρέπει όμως στο τέλος να είναι δυνατό να υποβληθεί μια πρόταση. Αλλιώς απλά θα έχουμε συναντήσεις ε, και θα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα καθυστερεί η συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αποτελεσματική συνεργασία στην ομάδα αυτή που θα συγκληθεί θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που να γίνονται σεβαστές και από τις δύο πλευρές. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα εντός των χωρών, ε, μεταξύ των χωρών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα μεταφορών και περιβάλλοντος. δεν ε, θα πρέπει να έχουμε έργα τα οποία οικονομικά να έχουν θετικό αντίκτυπο αλλά περιβαλλοντικά αρνητικό. Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή και ενισχυμένη συνεργασία. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας απλά να βρίσκει έναν εταίρο χωρίς να επιδιώκουμε μια λύση. αυτή τη στιγμή εντός ε, της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, ΜΟΥΒ αλλά και εντός της ΡΕΓΙΟ εξετάζουμε τα θέματα συνεκτικότητας. Είναι θέματα που συνδέονται και με το κλίμα. Η ΕΝΒΙ και η Γενική Διεύθυνση ΡΕΓΙΟ θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να υπάρχει περισσότερη συνοχή και επιτόπου. η εσωτερική ναυσιπλοεία και ιδιαίτερα οι σιδηρόδρομοι χρειάζονται συγχρηματοδότηση ύψους 30 με 35%. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων εδώ δεν είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο. Αυτό που θα δούμε και που βλέπουμε ήδη με τα προγράμματα που έχουν υποβληθεί είναι ότι στο Ευρωπαϊκό δίκτυο δεν έχουμε δώσει πολλή προτεραιότητα στους δρόμους, αλλά και εδώ υπάρχουν ανάγκες για επενδύσεις. Είναι λοιπόν εδώ ένα μέσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και στον ίδιο τον ΕΛΒΑ μπορούμε να επιδιώξουμε εταιρικέ σχέσεις. Γενικά η γύρω περιοχή σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων μας ενδιαφέρει. Αυτοί λοιπόν είναι τομείς τους οποίους ήδη έχουμε εντοπίσει στην ανάλυση που κάναμε. Όσον αφορά τις ερωτήσεις ε, του συναδέρφου Βιμ. Δεν είμαι τόσο κακός όσο λες. Σαφές είναι το εξής. Καθήκον μας είναι να εφαρμοστεί ο κανονισμός ΕΦΣΥ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτά που συμφώνησαν και αυτό που κάνουμε εδώ δεν είναι τίποτα καινούριο. Ξέρουμε από παλαιότερα πόσο δύσκολο είναι να εφαρμόσουν αυτά που έχουν συμφωνήσει. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τις προτεραιότητες από κοινού. Κατόπιν έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Μετά από όσα άκουσα ότι συνέβησαν ε, τη νύχτα, Μα ενδιαφέρει η σχέση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το Διευρωπαϊκό Δίκτυο. Θα πρέπει να μιλάμε όχι γενικά για μεταφορές, θα πρέπει να αναφερόμαστε στις προτεραιότητες. Εμείς αλλά και το Κοινοβούλιο μπορούμε να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τα θέματα αυτά, να θέτουμε ερωτήσεις, γνωρίζοντας βέβαια ότι ένα εργαλείο δεν μπορεί να ταιριάξει σε όλους. Συναντήθηκα στο λιμένα της Αθήνας, στον Πειραιά, ε, με τους Κινέζους. Και πρέπει να πω ότι ήταν ανοιχτή απέναντι σε εταιρικέ σχέσεις για περαιτέρω διασύνδεση του λιμένα. Ήταν διατεθειμένοι δηλαδή να συγχρηματοδοτήσουν. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, είναι καλό ή κακό αυτό. Εάν σεβαστούν τις προτεραιότητες του διευρωπαϊκού δικτύου, δεν θα πρέπει να εμποδίσουμε μια τέτοια χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτό είναι απλό θέμα. Και για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση. Η σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη προβλέπεται. Δεν φτάνει ο ίδιος ο διάδρομός μας μέχρι την Κωνσταντινούπολη, αλλά Η σύνδεση αυτή θα ενισχύσει την ε, μεταφορά εμπορευμάτων ε, και επιβατών. Έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν μια γωνιά της Βουλγαρίας όπου δεν γίνονται αρκετά και όπου απαιτείται βελτίωση της υποδομής για να έχουμε προστιθέμενη αξία. Αυτή λοιπόν η γραμμή νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθεί πάρα πολύ. Πάντως, ε, μας ενδιαφέρουν οι οικονομικές συνέπειες, μας ενδιαφέρει η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ετοιμαστείτε λοιπόν για, ένα δεύτερο, για μια δεύτερη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ματιέ Γκρός, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου. Κάτι ξέχασα και θα ήθελα να επενέσω την έκθεσή σου. προβλέπεται η γέφυρα στον Δούναβη ε, και αυτή τη γέφυρα την αναφέρω σε όλες τις ε, παρεμβάσεις μου διότι προβλέπεται για οδική μεταφορά, για το σιδηρόδρομο και για ποδηλατόδρομο. Μπορούμε λοιπόν έτσι τώρα να κλείσουμε τη σημερινή συνεδρία. Να ευχαριστήσω θερμά τον Ματιό Εγκρός και όλους εσάς. Πάντα χαιρόμαστε όταν έρχεται να μας δει. Η Λήξη τη συνεδρία.